Did you have for their for their longings and everything? Ladies and gentlemen, shall we get started? Have your seats. Καθίστε παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Να είστε ήσυχοι από τούδο και στο εξής παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούω συζητήσεις στην αίθουσα. Εκείνοι που θέλουν να κουβεντιάσουν, παρακαλώ ας βγουν από την αίθουσα για λίγο. Πρώτο σημείο είναι το σημείο 11. Αναπτυξιακές πτυχές όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα για γενετικές πηγές, πηγές γενετικού υλικού. Γνωμοδότηση της ΔΕΒΕ, που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Χέλμουτ Σόλτς είναι ο εισηγητής για σύνταξη της Η γνωμοδότησή μας θα πρέπει να αφορά εμπορικές πτυχές για το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να προχωρήσουμε σήμερα σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα σημαντικά αυτά θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε θέματα γενετικών πόρων και τις επιπτώσεις της μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρόκειται για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Η Κομισιόν στο μεταξύ έχει δημοσιεύσει σχέδιο κανονισμού και μετά από, τις, ε, από το πρωτόκολλο του Ναγκόγια. Ίσως λοιπόν εμείς να έχουμε μπροστά μας δύο κοινοβουλευτικές διαδικασίες για το θέμα αυτό. Και δεν είναι σαφές ακόμη ποια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα είναι αρμόδια επί της ουσίας. Υποθέτω όμως ότι λόγω του χαρακτήρα του θέματος η δική μας Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου δηλαδή θα συμμετέχει πάντως, θα αναμειγνύεται και στις δύο περιπτώσεις η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει την περίπλοκη κατάσταση που προκύπτουν από διάφορες ε, συμβάσεις, διεθνείς συμβάσεις, ε, συμφωνίες και ούτω καθεξής για την διανοητική διοκτησία για, τις, ε, τους γενετικούς πόρους. Θα πρέπει να συμβάλλουμε ώστε το θέμα να γίνει διαφανέστερο, πιο κατανοητό για τους καταναλωτές αλλά και για τους προμηθευτές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχει η Κομισιόν και σε επιτροπές εργασίας του, διεθνούς, ε, του παγκοσμίου μάλλον, ε, Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Ταυτόχρονα, το θέμα υπάγεται και στην ε, Σύμβαση περί βιοπικιλότητας και στο πρωτόκολλο του Ναγκόγια, το οποίο ακόμη δεν έχει όμως υπογραφεί και κυρωθεί από καμία χώρα μέλος. Ελπίζω το, το Κοινοβούλιο να μπορέσει να συζητήσει τα διάφορα αυτά θέματα στις διάφορες επιτροπές, αλλά βέβαια και η δική μας επιτροπή, έτσι ώστε να καταστεί σαφέστερο ότι πρέπει να κυρωθεί το πρωτόκολλο του Ναγκόγια στις διάφορες χώρες μέλη. Έχουμε και τα θέματα της συμφωνίας TRIPS, και επομένως δεν είναι εύκολο να υπάρξει μια συνεκτική λύση. Στην πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων θα ήθελα να θέσω ορισμένα θέματα και ιδίω ε, εμπορικά. Πρώτον, οι γενετικοί πόροι δεν μπορούν από τη φύση τους να είναι αντικείμενο άμεσο ε, ευρεσιτεχνιών συχνά βασίζονται σε παραδοσιακή γνώση. για τους γενετικούς πόρους ή για διάφορα μείγματα αυτών. Πώς όμως εμείς μπορούμε να βάλουμε την προσέγγιση αυτή μέσα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. θα πρέπει ο WIPO να αναλάβει την ηγετική ε, δράση ή θα πρέπει μάλλον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και τι μπορούμε να διδαχθούμε από την προσέγγιση άλλων χωρών σε σχέση με την παραδοσιακή γνώση που ανάγεται σε πέντε διαφορετικά είδη. Και εδώ παραθέτω από το πρωτόκολλο του Ναγκόγια το άρθρο 31 παράγραφος 1 που λέει ότι οι ηθαγενείς πληθυσμοί έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τον έλεγχο, να αναπτύξουν την παραδοσιακή τους κληρονομιά, γνώση και έκφραση, καθώς επίσης και τις εκφάνσεις της επιστήμης, πολιτισμού κλπ. και σε ό,τι αφορά ανθρώπινους και γενετικούς πόρους, καθώς και τις ιατρικές ή θεραπευτικές ιδιότητες ε, της Πανίδας και της Φλωρίδας, καθώς επίσης για παραδοσιακά, παραδοσιακές τελετές, παίγνια ή ε, άλλα σχετικά. Και να προστατεύεται η διανοητική διοκτησία επί της παραδοσιακής αυτής κληρονομιάς και των σχετικών της εκφάνσεων και εκφράσεων. Κάνω εγώ αυτή την παραπομπή εδώ διότι δίνει έτσι μια ε, συνολικότερη εικόνα του περί πρόκειται γιατί το πρωτόκολλο αυτό ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών όπου σημειώνεται ιδιαίτερα το πρόβλημα αυτό. Και ο αγώνας των θεγενών ε, ε, αυτών πληθυσμών είναι πώς να προστατεύσουν αυτή την κληρονομιά τους. Άλλο θέμα. Εάν υπάρχουν ωφελήματα, πλονεκτήματα που πρόκειται να μοιραστούν, Πώ θα εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι θαϊνεί πληθυσμοί θα λάβουν τα υλικά τα χρήματα. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι η αρχή της συνένεση μετά από πρώτερη ενημέρωση θα είναι εξασφαλισμένη. Και αναφέρομαι μόνο στο πρόβλημα εδώ των ηθαγενών πληθυσμών. Το ίδιο το θέμα όμως είναι ευρύτερο. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια νέα σφαίρα και πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Να λοιπόν ορισμένες από τις πτυχές που θα πρέπει να μας απασχολήσουν στη συζήτησή μας. Και αναμένω βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συνεργασία μαζί σας για να αναζητήσουμε τις καλύτερες λύσεις. Και επίσης απευθύνω χαιρετισμό στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, διότι αντιλαμβάνομαι ότι διαφορετικές γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν αναμειγνύονται στην εξέταση του θέματος. Έτσι λοιπόν σήμερα Κοντά μας είναι σήμερα η κυρία Μπάρμπαρα Νόκα από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, καθώς και άλλοι αρμόδιοι εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ονόματα στα πρακτικά. Uh, uh, καθώς και η Επιτροπή Προστασίας Υγείας και Καταναλωτών, Περιβάλλοντος, όλες αυτές οι Γενικές Διευθύνσεις Κομισιών συμμετέχουν και αναμειγνύονται, κάτι που κάνει το θέμα ακόμα πιο ενδιαφέρον. Το χρονοδιάγραμμα. 6 Νοεμβρίου, πρώτο σχέδιο. Ώστε να έχουμε τη δυνατότητα μαζί με τους κοιόδης να το συντάξουμε. Για τις τροπολογίες θα είναι 8 Νοεμβρίου. Και πάλι όμως προτείνω να κάνουμε πριν από αυτό μια συνεδρίαση για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τις διάφορες ιδέες. Και η ψηφοφορία στην Επιτροπή στις 28 Νοεμβρίου. Είναι σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, είμαι όμως αισιόδοξο ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και θα ακούσω βεβαίω με ενδιαφέρον τις άλλες απόψεις. Ευχαριστώ, Χέρμο Λοιπόν, εμείς μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο τις εμπορικές πτυχές του ζητήματος και όχι το πυρήνα του θέματος αυτό καθ' αυτό. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα μιλήσουν άλλα μέλη της Επιτροπής από τους ε, σκιώδεις, ο Κίστοφερ Φιόρνερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου πήρατε τις λέξεις από το στόμα μου, αυτά που θέλω να πω. Θα είναι πρόκληση αυτή να στιαθούμε μόνο στις εμπορικές πτυχές ε, μπορώ να βρω εκατομμύρια ενδιαφέροντα πράγματα προς συζήτηση. Και πού θα βάλει κανείς τη διαχωριστική γραμμή, τι συζητάμε και τι συζητάμε. Θα είναι δύσκολο να περιορίσουμε το πεδίο συζήτησης για να ασχοληθούμε αποκλειστικά με τα θέματα του διεθνούς εμπορίου. Θα είμαι λακωνικότατος. Εγώ ξεκινάω από το εξής που είναι σημαντικό δεν θα πρέπει να είναι άκαμπτη εφαρμογή της αρχής αυτή. Τόσο άκαμπτη ούτω ώστε να γνωρίσουμε τι δυνατότητες δημιουργούνται όσον αφορά του γενετικού πόρους. Πρέπει να εγγυηθούμε την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους για να έχουμε ιαδίποτε ωφέλη. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αυτό θα είναι άδικο. Όχι μόνο για διάφορους πολιτισμούς και λαούς με ιστορικές γνώσεις αλλά θα στερήσουμε και τα ωφέλη από τη χρήση αυτών γεωτικών πόρων από τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να είμαστε πολύ ανοιχτόμυαλοι. Σίγουρα αυτό θα κάνω. Όταν συζητούμε γύρω από τα θέματα αυτά στην Επιτροπή, έχουμε ένα περίεργο ιστορικό, αλλά ήθελα να το αφήσω πίσω μου. θα το κοιτάξουμε αργότερα. Εγώ δεν θα το κοίταζα από μια αμυντική θέση IPR των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα κινηθούμε, δεν θα πρέπει να αποκλίνουμε την πορεία μας πολύ. Διότι είναι από τους πιο δύσκολους τομείς όσον αφορά τα διανοητικά, τα πνευματικά δικαιώματα. Και θα είναι μεγάλη πρόκληση. Να συζητήσουμε το θέμα και εστιαζόμενοι μόνο στις εμπορικές πτυχές. Αυτό λέω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, ωραίο το αστείο στα αγγλικά. Copyright, left. Ε, λογοπαίγνιο. Κινούμαστε από τα δεξιά ή τα αριστερά τη ιδέα των μελλοντικών δικαιωμάτων. Δεν μεταφράσατε στα ελληνικά. Ο Χωσέ. Ή Χωσέ. Ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον και καθόλου εύκολο. Αν επικεντρωθούμε στην εμπορική πτυχή, αυτή είναι η αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, ε, τότε η έκθεση αυτή αποτελεί μια καινοτομία στα εμπορικά θέματα και στα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμφωνίες όπως ε, το πρωτόκολλο του Ναγκόγια είναι μια ισορροπημένη συμφωνία. Όμως τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο 27.3ε λέει ότι τα φυτά, τα ζώα, δεν πρέπει να μπαίνουν σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Εδώ όμως έχουμε και τους μικροοργανισμούς που μπορούν να μπουν σε πατέντα. Ε, ενώ τα φυτά όχι. Αν μεταπηθούν, ναι. Αν έχουν τύχη επεξεργασίας. Εδώ δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει ένα κενό. Θα έπρεπε να μπει εδώ μπροστά μας ε, το θέμα του συμφέροντος. Ποιος έχει να κερδίσει από αυτά. Ε, μια περιφέρεια, ένα κράτος, μια ομάδα ανθρώπων, μια περιοχή και η... μετά την εμπορία θα εξακολουθούν να κερδίζουν χρήματα οι αυτόχθονες οργανισμοί από τους οποίους ε, προέρχεται. Ξέρετε ότι με τους σπόρους είμαστε πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά την εμπορία των σπόρων. Είναι σημαντικό λοιπόν με την νομοθεσία να υπάρξουν κάποιες ε, λύσεις, αφού προηγουμένως βέβαια γνωρίζουμε πολύ καλά ε, τι ισχύει, είναι οι παραδόσεις και να λάβουμε υπόψη μας και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Μήπως αυτό θα ήταν μια λύση ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ε, στην περίπτωση που αποκαλύπτεται πάντα η πηγή. Είναι καινοτόμα πάντως ε, η ιδέα αυτή από πλευράς του εμπορίου και από πλευράς πνευματικής ιδιοκτησίας. Οπότε η Επιτροπή μας θα πρέπει να δουλέψει σκληρά για να συνδυάσει με κάθε λεπτομέρεια την εμπορία με τα πνευματικά δικαιώματα. Είμαστε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα, οπότε με τροπολογίες φαντάζομαι ότι θα διευκολύνουμε την κατάσταση για να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος που ζητάει το λόγο. Όχι. Ah, Αμέλια, and daughter from the Greens. Sorry. Η Αμέλια, εκπρόσωπος των Πρασίνων. Ευχαριστώ. The word. Um... Uh, λοιπόν, τα δικαιώματα των θαγενών χρησιμοποιούν παραδοσιακά φυτά και σπόρους και γνώση και γενετικούς σπόρους είναι κάτι αυταπόδεικτο. Αυτά τα δικαιώματα, πριν τα υπερασπιστούμε, δεν θα πρέπει να περιοριστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι σήμερα. Όταν ένα μονοπόλιο που παρεμβαίνει με το δικαίωμα των ηθαγενών να το κάνουν αυτό, βλέπουμε ότι τα πνευματικά δικαιώματα παραβιάζονται. Ταυτόχρονα, πολλέ στοιχείε του πρωτοκόλλου του Ναγκόγια και η Σύμβαση για την Βιοπικιλότητα, τη Γενετική, πρέπει να εξεταστούν προσεκτικότατα. Κάποιε αρχέ καθορίζονται με διαφορετικό τρόπο από τι άλλε διεθνεί συμφωνίε. Πολλέ βασικέ έννοιε και δικαιώματα δεν καθορίζονται επαρκώ. Αν μεγάλη προσοχή δεν δοθεί, υπάρχει ένα κίνδυνο για θέμητη και ασυνεπή εφαρμογή των κανόνων. Οι απαιτήσει τη Σύμβαση για την ε, βιολογική βιοπικιλότητα είναι αρκετά αυστηρέ. Η Σύμβαση και το πρωτόκολλο τη Ναγκόγια επικρίθηκαν διότι καθιστούν κάποιου τομεί έρευνα εκεί που κατοικούν κάποιοι ηθαγενεί ε, πιο δύσκολα λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Ποιο θα δώσει την άδεια για να χρησιμοποιηθούν τα δικαιώματα. Ποιο χορηγεί την πρόσβαση. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι αναπάντητα. The objectives of the οι στόχοι της σύμβασης για να, να αποτιμηθεί οικονομικά η βιοπικιλότητα ε, και να δίνονται ποσά στους σταγενείς δεν έχουν υλοποιηθεί, όμως οφείλεται κατά πολύ σε τεχνολογικές ε, διαδικασίες στο βιοτεχνολογικό τομέα, οπότε το πρωτόκολλο της Ναγκόγια δεν, μπορεί, δεν θα αλλάξει και πολλά πράγματα νομίζω. Το πρόβλημα της βιοπειρατείας, όταν αυτή είναι πραγματική, είναι ένα πρόβλημα πολλών πνευματικών δικαιωμάτων τυπικά διπλωμάτων ευστεχνίας. Αν υπάρχουν πάρα πολλά πνευματικά δικαιώματα, ε, το πρόβλημα αυτό δεν θα επιληθεί αν προσθέσουμε και άλλα πνευματικά δικαιώματα στο μείγμα. Πιστεύω στα δικαιώματα, το δικαίωμα της ελευθερίας για τους λαούς. Όχι να αποκλείονται οι άλλοι όμως από τη χρήση ή τον επιμερισμό της γνώσης. Χρειάζεται πιο αποτελεσματική και ισότιμη λύση για την βιοπειρατεία οι παραδοσιακέ γνώσει και οι παραδοσιακοί γενετικοί πόροι να εξαιρεθούν από τα πνευματικά δικαιώματα και την τεχνία. Έτσι θα μειωθεί το κόστος συναλλαγών και θα εξασφαλίζεται ε, ισότιμη πρόσβαση και ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και αυτή είναι η θέση πολλών στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες των ιδίων των λαών που προσπαθεί να βοηθήσει η, ε, η σύμβαση αυτή. Έχουμε και θετικέ, πολύ θετικέ εμπειρίε όσον αφορά την αποκάλυψη στοιχείων και σχόλια όσον αφορά για τα πορίσματα τη γενετική έρευνα και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, πιστεύω, στην γνωμοδότηση. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Α ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τι διαφορετικέ γενικέ διευθύνσει εδώ. Η Μπάρμπαρα Νόρκρο από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε όλους. Νομίζω ότι είναι η αρχή μιας πολύ ενδιαφέρουσας περίοδου όπου το Κοινοβούλιο βεβαίως θα συμμετάσχει πλήρως στις συζητήσεις για την πρόταση για την εφαρμογή του πρωτοκόλου της Ναγκόγια. Υπάρχουν πολλές γενικές διευθύνσεις που συμμετέχουν. Βλέπετε κάποιους εκπροσώπους αυτών εδώ σήμερα. Αυτό που θα σας έλεγα πέρα από τις επιπλοκές που φοβούνται κάποιοι ότι εστέ βέβαιοι ότι όλοι κοπηλατούμε προς την ίδια κατεύθυνση και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας μαζί, το ταχύτερο δυνατόν. Από πλευράς Γενικής Διευθύνσεω Εμπορίου νομίζω ότι η κατάσταση είναι η εξής. Η Σύμβαση για τη Βιοπικιλότητα και πώς σχετίζεται αυτή με τη Συμφωνία TRIPS ε, είναι κάτι που συζητείται επί σειρά ετών. Ε, βεβαίως ακούμε, πηγαίνουμε στον ΠΟΕ, και παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα όσον αφορά τη Σύμβαση για τη Βιοπικιλότητα και νομίζω ότι υπάρχει γενική συμφωνία ότι οι συμφωνίες οι δύο τρίψ του ΠΟΕ και η Σύμβαση για τη Βιοπικιλότητα πρέπει να αλληλοϊποστηρίζονται. Αλλά επίση υπάρχει συμφωνία ότι όσον έχουμε κάτι καινούργιο στη Σύμβαση για την Επικοινότητα υπό τη μορφή του πρωτοκόλου τη Ναγκόγια, στον ΠΟΕ θα πρέπει να περιμένουμε να περιμένουμε του το πρωτόκολλο της Ναγκόγια να τεθεί σε ισχύ, σωστά. Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι συμβαίνει στην WIPO, διότι εκεί συζητούν ε, πιο ουσιαστικά ζητήματα περί γενετικών πόρων και παραδοσιακής γνώσης. Ακούμε, αφού κραζόμαστε, αλλά περιμένουμε επίσης. Και πράγματι δεν θέλουμε, κύριε Άντες, τότε να επιφέρουμε περαιτέρω σύγχυση. Είναι καλύτερα να περιμένουμε οι συζητήσεις στα δύο προανθαφερθέντα βήματα να ολοκληρωθούν πριν δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς στα πλαίσια της συμφωνίας TRIPS. Καλό να απομακρυνθούμε από συναισθηματική συζήτηση για τα πνευματικά δικαιώματα το πρωτόκολλο της Ναγκόγια πρέπει να ειδωθεί ως κάτι άκρος εποφέλες. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Αυτές οι θαγενείς κοινότητες θα έχουν δυνατότητα να πούνε ναι ή όχι, αν θέλουν γενετική του σπόροι να χρησιμοποιηθούν ή όχι. used, will... Εάν ναι, επιτρέψουν να χρησιμοποιηθούν, θα έχουν τη δυνατότητα να πούνε υπό ποιους όρους θα χρησιμοποιούνται. Και όποιο θέλει να χρησιμοποιήσει οσδήποτε από αυτού του γενετικού πόρου θα πρέπει να πάρει την άδειά του και θα πρέπει να είναι διαφανή και επίσημη διαδικασία. Ενθαρρύνω λοιπόν την Επιτροπή Ίντερ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεργαστούν καλά με τι άλλε επιτροπέ και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά. Όλοι θέλουμε αυτέ οι θαγενεί κοινότητε να ωφεληθούν στο μέτρο του δυνατού από του ίδιου γενετικού του πόρου. Σα ευχαριστούμε. Έχω δύο ονόματα από την Γενική Διεύθυνση Αγοράς. Μάρκτα. ποιος ε, θα μιλήσει εκ μέρους, ο Μάικλ Πράιερ ή ο Αλφόνσο Κάγιες Σάνσεθ. Καλημέρα. Αλφόνσο Κάγιες ονομάζομαι από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς από την, το τμήμα βιομηχανικής ε, ιδιοκτησία. Θέλω να σας ε, μιλήσω λοιπόν για το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησία. Εδώ και αρκετά χρόνια μέχρι σήμερα στην WIPO συζητάμε ορισμό. Πώς να ρυθμίσουμε τις παραδοσιακές γνώσεις και τους γενετικούς πόρους και ό,τι έχει να κάνει με παραδοσιακές ε, συνήθειες, με έθιμα. Αποφασίστηκε για την επόμενη χρονιά ότι θα συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα θέματα Υπάρχουν ε, τρία σχέδια κειμένου και για τα έθιμα και για τις παραδοσιακές συνήθειες και για τις ε, παραδοσιακές γνώσεις και τον επόμενο χρόνο θα υποβάλουμε ένα τελικό κείμενο και θα αποφασιστεί κατά πόσο θα γίνει και μια διπλωματική διάσκεψη στο μέλλον ή όχι. Εξαρτάται πόσο θα έχουμε προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις αυτές. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πιστεύουμε αυτό, οποιοδήποτε μέτρο ή σύστημα δημιουργηθεί σε αυτό το τομέα πρέπει να γίνει σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι η γνώμη μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε κοινή θέση για την ε, αποκάλυψη της ε, πηγής όταν ε, μιλάμε για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας από το 2005. Το 2005 δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 25 χώρες μέλη συμφώνησε κοινή θέση για το πώς να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό της αποκάλυψης ε, των γενετικών ε, πηγών στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αυτή την πρόταση λοιπόν την πήγαμε και στο ΟΑΠΟ και στον ΠΟΕ. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν αυτή τη θέση έχουν. Επίσης, όπως ακούσαμε και σήμερα το πρωί, υπάρχει και οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αναφέρεται στα διπλώματα βρεσιτεχνίας για την βιοπικιλότητα. Αυτά είχα να σχολιάσω στον τομέα της βιομηχανικής ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και ό,τι άλλο θέλετε ευχαρίστως να σα απαντήσουμε για τις νομικές πτυχές, τις πρακτικές πτυχές ή οτιδήποτε έχει να κάνει με το IPR, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οτιδήποτε άλλο. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ τώρα. έχω κυρίες. Η κυρία Μάνα Κόλπη, η κυρία Κλεμόνισου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω κάποια σχόλια εκ μέρους της ΑΝΚΟ. Είμαι, ονομάζομαι Κάπερκοφ και έχω και εγώ ως θέμα τα βιομηχανικά υλικά. Μιλάμε τώρα για την κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Τώρα μιλάμε για τα φυτά που είναι κάτι πιο λεπτό από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, γενικά, γιατί υπάρχουν εδώ πέρα εξαιρέσει. Δεν καλύπτονται και δεν προστατεύονται όλες οι ποικιλίε. Αν λοιπόν δεν προστατεύονται οι ποικιλίε, καταλαβαίνετε ότι μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν στις καλλιέργειες. Ένας άλλος ο τομέας ε, είναι, με τον οποίο ασχολούμαστε είναι η γενετική πόρη. Νομίζω ότι εδώ όλοι θέλουμε να πετύχουμε τους ε, ίδιους στόχους, τους στόχους της ε, έκθεσης. Το πρωτόκολλο Ναγκόγια, το οποίο καθορίζει τη διαδικασία σε διεθνές επίπεδο για τα κέρδη και την πρόσβαση στα κέρδη και την κατανομή των κερδών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η ΣΑΝΚΟ είναι υπεύθυνη και για την Διεθνή Συμφωνία όσον ε, αφορά τους γενετικούς πόρους για τα τρόφιμα. Πολλά χρόνια έχουμε δουλέψει λοιπόν μέσα σε αυτό το ε, πολυμερές ε, σύστημα. Πιστεύουμε ότι μπορεί να βελτιθεί ακόμα περισσότερο τώρα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο εισηγητής πάλι για να μας πει τα σχόλιά του. Είναι σαφές ήδη ότι υπάρχουν πολλές πτυχές εδώ που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην γνωμοδότησή μας. Δεν θα προσθέσω άλλα ερωτήματα, ούτε θα καταλήξω σε συμπεράσματα εφόσον είμαστε σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Συμφωνώ πάντως ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις πτυχές που έχουν να κάνουν με το εμπόριο. Αλλά βλέπετε το εμπόριο καλύπτει και άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη η οποία πρέπει να οριστεί πολύ συγκεκριμένα. ο ορισμός που προτείνεται έχει κοινή αποδοχή πιστεύω για τα δικαιώματα πραγματικής ιδιοκτησίας σε γενετικούς πόρους, οπότε πιστεύω ότι μπορεί αυτό να μας βοηθήσει και έτσι να καταλήξουμε σε, με τη γνωμοδότησή μας σε μια πιο συγκεκριμένη άποψη πάνω στο θέμα αυτό. Ε, περιμένω ακόμα τους συναδέρφους ό,τι σχόλια έχουν να κάνουν σε αυτό το πρώτο σχέδιο μέχρι αρχές Νοεμβρίου είμαι στη διάθεσή σας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, αυτή, ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε για αυτό το θέμα. Το επόμενο είναι, ή στις 6 Νοεμβρίου θα ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Και ερχόμαστε τώρα στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 12. Έχουμε παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά τις προσχωρήσεις των ΠΟΕ. Όπως γνωρίζετε ήδη έχουμε Λάος, Τατζικιστάν. Εδώ θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Κάρλος Χιμένες. Σε εσάς θα δώσω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους σας εδώ. Ο Πρόεδρος διακόπτη. Κάνετε πάρα πολύ φασαρία σε αυτή την αίθουσα. Χρειάζεται να το επαναλαμβάνω κάθε φορά, σε κάθε συνεδρίαση ξανά και ξανά, ότι δεν μπορώ να δεχτώ πηγαδάκια μέσα στην αίθουσα. Παρακαλώ κύριε σε Ευχαριστώ και πάλι πρόεδρε και πάλι καλημέρα σε όλους εδώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την προσχώρηση στον ΠΟΕ. Θέλω να αναφέρω ότι το 2012 ήταν μια πολύ παραγωγική χρονιά. Είχαμε το Μαυροβούνι, τη Σαμό και το Μπενό που προσχώρησαν στον οργανισμό. Τα μέλη που έχουν προσχωρήσει είναι πολύ περισσότεροι από αυτοί που έχουν προσχωρήσει, πολύ περισσότεροι από αυτούς που περιμένουν να ενταχθούν. 29 έχουν προσχωρήσει, 26 περιμένουν να ενταχθούν. Γίνεται λοιπόν, ε, υπάρχει πρόοδος για τις αναπτυσσόμενες χώρες. αναθεωρήθηκαν οι καθοδητήρες γραμμές για την προσχώρηση των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών στον ΠΟΕ. Ετέθηκαν διάφορα, διάφορες προϋποθέσεις, διάφορα όρια για την προσχώρησή τους, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά, κυρίως και για τις μεταβατικές περιόδους. Όμως, λιγότερο θετικό είναι η στάση κάποιων χωρών που πρόσφατα προσχώρησαν και οι οποίες δεν διευκολύνουν την κατάσταση γιατί δυσκολεύουν την προσχώρηση άλλων που μέχρι τώρα ήταν φιλικές τους χώρες. Η Ουκρανία, για παράδειγμα, καθυστερεί το Μαυροβούνι. Και με το Λάος και την Ιεμένη δυσκολεύονται πολύ οι διαπραγματεύσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν δυσκολίες και για την περίπτωση του Τατζικιστάν, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα και να ενταχθεί στον ΠΟΕ. Όπως είπα, υπάρχουν, ε, διάφορες, υπάρχουν αυτές οι δύο τάσεις, ε, η μία που διευκολύνει τις προσχωρήσεις και η άλλη που τις εμποδίζει, τις δυσκολεύει. Το Λάος και το Τατζικιστάν πάντως βρίσκονται πιο κοντά στην προσχώρηση. Σας είπα ότι η Ουκρανία καθυστερεί κάπως ε, τις προσχωρήσεις, αλλά τώρα πάντως όλο το σχέδιο πακέτου έχει εγκριθεί στην τελευταία ομάδα εργασίας 28 Σεπτεμβρίου. Η προσχώρηση του Λάος λοιπόν θα υποβληθεί στο Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕΣ στις 26 Οκτωβρίου σε μια ειδική δηλαδή έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Όλες οι διαδικασίες εσωτερικές έχουν ολοκληρωθεί, η απόφαση έχει πάει ήδη στο Συμβούλιο και ελπίζουμε ότι θα εγκριθεί πολύ γρήγορα ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει και εκείνη τη συνένεσή της στο Γενικό Συμβούλιο. Όσον αφορά το Τατζικιστάν, Ήμουνα στην ε, Γενέβη την τρίτη που μας πέρασε. Η προπαρασκευαστική δουλειά έχει ολοκληρωθεί για να υιοθετηθεί στη συνεδρίαση της, ε, για να, στις 9 ε, Οκτωβρίου, δηλαδή την ίδια μέρα την ομάδα εργασίας, προκειμένου να εγκριθεί εκεί. Όλοι θέλανε να συμφωνήσουν και η Ρωσία Μάλλον η Ρωσία έκανε, όμως έβαλε ένα διαδικαστικό θέμα. Είπε ότι χρειάζεται τέσσερις εβδομάδες για να μελετήσει τα έγγραφα. Αγνώντα ότι τα έγγραφα ήταν στη διάθεσή τους από τις 20 Αυγούστου σε κάποια άλλη μορφή, Οπότε τώρα γι' αυτό καθυστέρησε το πράγμα και γι' αυτό πάει στις 26 Οκτωβρίου. Αν τώρα όλα αυτά τα διαδικαστικά λυθούν, ελπίζουμε να έχουμε την τελική έγκριση στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ που θα γίνει 11 και 12 Δεκεμβρίου το τελευταίο για φέτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ξέρετε ότι έχει κάνει όλη την προπαρασκευαστική δουλειά και θα υποβάλουμε την, ε, το σχέδιο απόφασης και αν εγκρίνει το Γενικό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτοιμη να δώσει τη δικιά της ε, συνένεση. Στην περίπτωση της Ιεμένης υπάρχει επίσης πρόοδος, αλλά η Ουκρανία καθυστερεί τις ε, διαπραγματεύσεις. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε νέα ημερομηνία για την ομάδα εργασίας προκειμένου να εγκρίνει το πακέτο και μετά να προχωρήσουμε στην γενικότερη έγκριση. Άλλες προσχωρήσεις ε, προοδεύουν, όχι για το εγγύης μέλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει του χρόνου θα έχουμε πιστεύω καλά νέα για το Καζακστάν όπου δουλέψαμε την προηγούμενη εβδομάδα στην Γενέβη πολύ εντατικά. Έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος, αλλά υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα, αν όχι και τρία που πρέπει να λυθούν. Το πρώτο είναι ότι η νομοθεσία του Καζακστάν περιλαμβάνει πολλές απαιτήσει όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, την ενέργεια για όλες τις επιχειρήσεις που ανήκουν στο κράτος. Είναι δηλαδή τοπικές προϋποθέσεις οι οποίες είναι σύμβατες όμως με το καθεστώς του ΠΟΕ. Το Καζακστάν το αναγνωρίζει αυτό και θα προσπαθήσει να πετύχει μεταβατικές περιόδους για να συμμορφωθεί με τα TRIMS. Αυτή θα καλύψει την περίοδο μέχρι να λήξουν οι συμβάσεις αυτές που έχει σε τοπικό επίπεδο το Καζακστάν. Μέχρι το 2042 για παράδειγμα. Βέβαια τέτοια πρόταση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και καταλαβαίνετε ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ τι διαπραγματεύσει. Η δεύτερη δυσκολία για τις διαπραγματεύσεις μας αυτές έχει να κάνει με τους δασμούς που ήδη έχει διαπραγματευτεί το Καζακστάν με πολλά μέλη του ΠΟΕ προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τους δασμούς της Τελωνιακής ε, Ένωσης, από με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Η διαδικασία αυτή θα είναι περίπλοκη. Θυμίζει λιγάκι αυτό που ε, πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά που προχωράει σε διεύρυνση. Άλλες δύο προσχωρήσεις τώρα υπάρχουν που θα προχωρήσουν γρήγορα φαντάζομαι στο μέλλον, Βαλκανικές χώρες, Σερβία και Βοσνία. Εδώ οι διαπραγματεύσεις έχουν προχωρήσει πολύ. Από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτό που προσπαθούμε μάλιστα να κάνουμε είναι να συντονιστούμε μαζί τους όσο γίνεται καλύτερα για τις θέσεις μας. Στα πλαίσια της διεύρυνσης μάλιστα έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να έχουν υιοθετήσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οπότε ό,τι και να κάνουν στη διαδικασία προσχώρησής τους δεν θα πρέπει να αντιβαίνει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ναι. Αυτά έχω να σας πω. Από εκεί και πέρα αν έχετε ερωτήσεις, σχόλια, ευχαριστώ να απαντήσουμε. Σας ευχαριστώ. Πάμε στα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Άκουσα αυτά που λέγατε. Χτες, μάλιστα, είχαμε μια συνεδρίαση της ε, ομάδας ε, παρακολούθησης ε, για τη Ρωσία. Τέσσερα μέλη που είναι εδώ παρόντα ήταν σε αυτή τη συνεδρίαση. Εγώ έφυγα πολύ ανήσυχο χθε για τη θέση της Ρωσίας. Και μας λέτε τώρα ουσιαστικά ότι η Ρωσία θα είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα για κάποιες από τις χώρες που θα μπουν στον ΠΟΕ. Θα είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όπως το περιγράψατε και διαστανόμαστε. θα προσπαθήσει να μπλοκάρει διάφορες χώρες να μπουν. Πρώην δηλαδή χώρες που ήταν ε, σοβιετικοί δορυφόροι θα προσπαθεί να μπλοκάρει την είσοδό τους ε, στον ΠΟΕ, η Ρωσία. Κέλλερ, κύριε Κέλλερ, ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια του γύρου της Ντόχα, οι αναπτυσσόμενες χώρες ζητούσαν οι κανόνες για την προσχώρηση στον ΠΟΕ να αλλάξουν για να διευκολυνθεί η πρόσβασή του στον ΠΟΕ, η προσχώρησή του στον ΠΟΕ. Από αυτά που ακούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στηρίζει αυτά τα αιτήματα. Αν δούμε όμως τις λεπτομέρειες, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους βασικούς φορείς που ζητάει περισσότερες φιλελευθεροποίησεις εκαπιστομής τα, οι νέε χώρε θα πρέπει να καταργήσουν όλου του εξαγωγικού περιορισμού και να δεσμευτούν να μην εισαγάγουν νέες εξαγωγικές, νέους εξαγωγικούς περιορισμούς στο μέλλον. Αυτή είναι μία απέτηση. Και θα πρέπει να έχει συμμόρφωση με τους κανόνες ΠΟΕ. Ζητάει ΠΟΕ συν, κανόνες ΠΟΕ συν για τις νέες χώρες. Παρόλο που υπάρχουν σαφείς κανόνες γιατί δεν χρειαζόταν συμπληρωματικοί κανόνες, γιατί δυσκολεύονται οι χώρες, κυρίως οι αναπτυσσόμενες έτσι να προσχωρήσουν. Ερώτηση. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποστηρίζεται το αίτημα των αναπτυσσόμενων χωρών να διευκολυνθεί η προσχώρησή τους ή ζητάτε από όλα τα νέα μέλη του ΠΟΕ περισσότερες α, δεσμεύσεις από ό,τι τις συνηθισμένες. Θα σταματήσετε να επιμένετε να καταργηθούν τώρα όλοι οι εξαγωγικοί περιορισμοί που επιβάλλουν αυτές οι χώρες και τώρα και στο μέλλον, οι νέες, οι αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν υπάρχει άλλο να πάει το λόγο, λέει ο πρόεδρος, από ό,τι βλέπω. Έχω και εγώ ερώτηση. Μου λέει ένα σημείωμα εδώ ότι καλέ, πολλές ε, χώρες ε, στην Κεντρική Ασία και λοιπά που δεν έχουν προσβαση στη θάλασσα όπως είναι το Καζακστάν, το Τατζικιστάν. Συναντήθηκα στην Άλμα Άτα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Πάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you. I Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που ετέθησαν τα ερωτήματα. Η θέση της Ρωσίας. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η Ρωσία δεν αισθάνεται άνετα όταν οι χώρες της ευρύτερης περιοχής που προσχωρούν στην Τελωνιακή Ένωση ή στην Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που θα υπονόμευαν ενδεχομένως αυτά που προσπαθούν να πετύχουν σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή, κανένα το πω, είναι υπονομεύουν τι σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό ίσως δημιουργήσει δυσκολίες όταν αυτές οι χώρες όπως το Τατζικιστάν είναι αποφασισμένες να προσχωρήσουν στον ΠΟΕ και έθεσαν ως προτεραιότητα να προσχωρήσουν στον ΠΟΕ πιο πάνω από ότι να συμμετάσχουν στο περιφερειακό μόρφωμα. Την Τρίτη το είδαμε αυτό όταν διακεκριμένος ε, ε, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι η Ρωσία με διαδικαστικούς τρόπους μπλοκάρει την προσχώρηση του Τατζικιστάν και ο Ρώσος εκπρόσωπος προσβλήθηκε και είπε δεν μπλοκάρω τίποτα, δεν μου αρέσουν αυτοί οι πενιγμοί, ζητώ απλώς να γίνει σεβαστή η όλη διαδικασία που χρειάζεται τέσσερις εβδομάδες. Ε, ε, έχει σταθεροποιηθεί το όλο πακέτο από ό,τι καταλαβαίνουμε και σε τέσσερις εβδομάδες αν υπάρχει μπλοκάρισμα θα πρέπει να θέσει το ζήτημα η Ρωσία ξεκάθαρα στα υπόλοιπα μέλη. Τώρα για τις χώρες που θέλουν να προσχωρήσουν και τους εξαγωγικούς δασμούς. Διευκρίνηση. Μετά την 8η Υπουργική Διάσκεψη αποφασίστηκε οι κατευθυντήριες γραμμές να αναθεωρηθούν για την προσχώρηση των λιγότερων επιτυγμένων χωρών. είναι προσανατολισμοί, κατευθύνες γραμμές. Δεν υπάρχει πλήρης ακαμψία. Ζητείται αυτό περιορισμό όσον αφορά τις απαιτήσει που τίθενται για τις λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε. Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες τώρα που περιμένουν να προσχωρήσουν στον ΠΟΕ, αυτές οι κατευθυντές γραμμές δεν ισχύουν. Διεξάγονται διμερείς ε, διαπραγματεύσεις. Και ακολουθείται μεταρρυθμιστική διαδικασία και ένταξη στο πολυμερές σύστημα εμπορίου. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ θεωρεί ότι οι εξαγωγικές επιδοτήσεις στρεβλώνουν το εμπόριο και θέλουμε να εξαλειφθούν ή να μειωθούν ουσιαστικά. Και αυτό το ζητάμε στις διαπραγματεύσεις. Αυτή είναι η να μειωθουν ουσιαστικα και αυτο το ζηταμε στι διαπραγματευσει αυτη ειναι η πολιτικη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά μπορώ να πω επ' αυτού. Πρέπει να κάνουμε, κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και επαναλαμβάνουν τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι εξαγωγικέ επιδόσει τρευλώνουν το εμπόριο και θα πρέπει ε, να μειωθούν. Όσον αφορά τις χώρες ε, που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα, είναι μια διαδικασία που δεν είναι του ΠΟΕ, αλλά της UNCTAD. Και λαμβάνουμε υπόψη τις πτυχές τις ιδιαίτερες για αυτές τις χώρες. Ήμουν στη Γενέβη την περασμένη εβδομάδα, στι συζητήσεις. Και το Καζακστάν και το Τζικιστάν δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και αυτό αναφέρθηκε επανειλημμένα για να ληφθεί υπόψη το αίτημά τους. Θέλουν επιδοτήσεις για να αντισταθμιστούν τα μεταφορικά έξοδα κλπ. Το έχουμε όλοι υπόψη αυτό και θα εξεταστεί. Δεν υπάρχει όμως απόφαση το ΠΟΕ για τις χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στη θάλασσα. Από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω. Φρανσίσκα Κέλλερ, ζήτησε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Ε, λυπούμε. Ίσως να παρεξηγήσετε την ερώτησή μου. Ε, μίλαγα για τους εξαγωγικούς περιορισμούς, όχι τις επιδοτήσεις. Ε, είναι, είναι κάπως διαφορετικό αυτό και σε αυτό αν μπορούσαμε να απαντήσετε ο εκπρόσωπο της Κομισιόν, χέρι με χέρι πάνε αυτά. Εξαγωγικοί περιορισμοί θεωρούνται ότι στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και αν γνωρίζω καλά όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και όταν γίνεται αυτή η συζητήση στον τομέα αυτό, στην αρμόδια γενική διεύθυνση, θεωρείται ότι αυτοί οι περιορισμοί έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα για τη διατροφή του πληθυσμού στον κόσμο ε, πολύ συχνά. Ευχαριστώ. Καλώς. Αυτά είχαμε να πούμε πριν έρθει η ώρα των ψηφοφοριών. Ας κάνουμε διακοπή δύο λεπτών, ούτως ώστε τα μέλη της Επιτροπής μας να μπορέσουν να προσέλθουν. Ετοιμαστείτε, ε. κάρτες ψηφοφορίες κλπ. Κατάλογο ψηφοφοριών κλπ. Are Let's move on. Voting time. First item... Λοιπόν, πρώτο σημείο. Διαδικαστική απόφαση. Για τον κανονισμό για την πρόσβαση στην αγορά, όπως αποκαλείται. Να ξεκινήσουμε να πραγματεύσουμε το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να φτάσουμε στη συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση. Διότι οθετήσαμε τη θέση μας στην πρώτη ανάγνωση στην Ολομέλεια πριν από δύο εβδομάδες περίπου. Ο David Μάρτιν, ο εισηγητής μας, έχει κάτι να μας πει. David Μάρτιν. Κανονισμός για πρόσβαση στην αγορά. Διαδικαστική απόφαση. Τι πρέπει να κάνουμε από τούδε και στο εξή. Απεριμένουμε είναι η απάντηση. Το Συμβούλιο ακολουθεί διαδικασία δεύτερης ανάγνωσης, να περιμένουμε να τελειώσει το Συμβούλιο και να κάνουμε τα δέοντα, αν προχωρήσουν γρήγορα, μπορούμε ίσως τον Νοέμβριο στη συνεδρίασή μας να αποφασίσουμε, αλλά πρέπει να περιμένουμε πόσο γρήγορα θα κινηθούν αυτοί. Εντάξει, λέει ο Πρόεδρος, ε, συμφωνείτε να αναβάλουμε το θέμα αυτό. Καμία αντίρρηση. 14, σημείο 14. Δασμολογικές ποσοστές περιπτώσει εξαγωγέ ξυλία από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χορήγηση δεσμολογικών ποσοστώσεων. Ηλεκτρονική ψηφοφορία που ξεκινάει. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 24 ψήφοι υπέρ, 2 αποχές, καμία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια λοιπόν. στη συγκήτρια. 15 ενωσιακός τελωνιακός κώδικας ε, της κυρίας Μοσκαρντίνη. Η Κριστιανά Μοσκαρντίνη είναι η συγκήτρια. Στις τροπολογίες 3 και 15 έχει ζητηθεί ξεχωριστή ψηφοφορία. 3 υπέρ, τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ. Αυτό είπα στην αρχή ότι θα ψηφίσουμε χωριστά, σας το είπα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο ηλεκτρονικός έλεγχος στην τροπολογία 5. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. 16. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 μάλλον 20 λέει ο πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τι είπατε έλεγχος για την 6 ηλεκτρονικός έλεγχος της 6 ξεκινάει πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε 25 ψήφοι υπέρ. Ήταν ε, μικρή διαφορά των ψήφων, λέει χαριτολογώντας ο πρόεδρος. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται έλεγχος ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 9 άρχεται η ψηφοφορία για την 9 πέρας ψηφοφορία. εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 και 13. Α, 12. Ξεχωριστά λοιπόν. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 2. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. «26 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, καμία ψήφος εναντίον» πλήρης η επιτυχία της κυρίας Μουσκαρντίνη. Συγχαρητήρια. Πάμε... Στο σημείο 16 Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες Ο πρόεδρος είναι ο εισηγητής Τροπολογία 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 Ας προχωρήσουμε στη συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για την 49 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Απερίφθη. Τροπολογία 15 υπέρ. 50 μα συγγνώμη εποχές. Εγκρίνεται. 50, όχι, γιατί είπε 15. 50. Εγκρίθηκε η 50 και όχι 15. 50. 53 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 54 υπέρ, Προφορική τροπολογία. Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Ο κ. Ρόβολ μου ζήτησε να υποβάλω προφορική τροπολογία. Το διευρυμένη enhanced ε, να αφαιρεθεί δύο φορές από την τροπολογία 54. Το enhanced, δύο φορές. Αντίρρηση για την προφορική τροπολογία, αλλά πρόεδρο, όχι, καμία αντίρρηση. Θα ψηφιστεί ως ετροποποίηθη προφορικό. υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 55 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες 58, 59, 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Έλεγχος τις τροπολογίες 58, 59 και 60. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 69 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απερίφθη 68 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές Α, απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος για την 73. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 74 και 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αν δεν κάνω λάθος, σας γίνει έλεγχος για την 76, ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 83 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την τροπολογία 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Όχι. Συγγνώμη. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 έτσι δεν είναι. 98 συμβατή με τη συμβαστική 8 98 υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος ας γίνει έλεγχος για την 98 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε Συμβαστική 9. Υπέρ. Μου λένε ότι πρέπει να ψηφίσουμε την 100. Στην 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 100. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία. Συμβιβαστική 9. Compromise 9 in favor. Συμβαστική 9 υπέρ. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έλεγχος για την 107. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. Τροπολογία 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ο κ. Κασπάρη. Να ελεγχθεί αν η τροπολογία μου 101 α, καταπίπτει. Η συμβαστική 8 εγκρίνεται. Μπορείτε να ελέγξετε τι γίνεται με την δική μου τροπολογία μέχρι ότου γίνει η τελική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Γραμματεία. Για την τροπολογία 101, λέει ο Πρόεδρος. Μου λέγουν ότι η διατύπωση εμπεριέχεται στη συμβιβαστική που ήδη ψηφίστηκε. Και εμείς έχουμε το ίδιο ερώτημα για την 110. Ίσως το έξυπνο είναι να ψηφίσουμε και ελέγχουμε μετά, για να είμαστε σίγουροι. Αν θέλετε, λέει ο Πρόεδρος. Πάμε πίσω λοιπόν. Επιστρέφουμε στην τροπολογία 101. Πάμε πίσω λοιπόν. Στην 101, τροπολογία 1, 101 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε κανονικά την ψηφοφορία μας. Πάμε στον κατάλογο. Συμβιβαστική 10. Την 110 μπορούμε να την ελέγξουμε παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Ας ελέγξουμε την 110. Άρχεται η ψηφοφορία για την 110. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 έλεγχος για την 116 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Απερίφθη. Almost a draw. Σχεδόν ε, ισοψηφία, λέει ο πρόεδρο. 117 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται, δεύτερο τμήμα υπέρ. Α, καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 120 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ενεκρίθη. Τροπολογία 122 υπέρ 122 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται 123 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογικές σκέψεις. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 10 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 22 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ έλεγχο 26 Ηλεκτρονικό έλεγχος για την 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ενεκρίθη. 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αιτιολογικές αναφορές 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έκον 7 έκον 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έκον 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αν δεν κάνω λάθος σας ελέγξουμε έκον 8 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε λοιπόν ΥΜΚΟ 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. ΥΜΚΟ 5 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είμαι σίγουρος. Ας ελέγξουμε. Πρώτο τμήμα της ΙΜΚΟ 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. εγκρίθηκε δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απερίφθη ΙΜΚΟ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 7 υπέρ κατά περίφθη ΙΜΚΟ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και ΙΜΚΟ 9 α καταπίπτει τραν μεταφορών Τραν 2 Τραν 2 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Τραν 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τραν 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Για την Τραν 4 ας γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορία. Απερίφθη. Σχεδόν ισοψηφία λέει πάλι ο πρόεδρο. Ψηφίζουμε το σχέδιο εκθέσεως ω ετροποποίηθη η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίθηκε 24 ψήφοι υπέρ, 4 ψήφοι κατά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ σου συνέβαλαν στη βελτίωση της έκθεσης μου. Να σας πω ότι η ένδειξή μου να καταψηφιστούν κάποιες τροπολογίες δεν σχετιζόταν με την ουσία. Σε κάποιες περιπτώσεις θα συμφωνούσα με την ουσία των τροπολογιών, αλλά θεώρησα ότι ήταν εκτός πεδίου πολύ λεπτομερής, θα υπερφόρτωναν την έκθεση και νομίζω ότι αυτή η έκθεση που είναι η πρώτη έκθεση επ' αυτού του σημαντικότατου ζητήματος θα έπρεπε να είναι σαφής, αυτοπεριορισμένη, με σαφές ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Item 17. Τώρα ακολουθεί το θέμα υπαριθμό 17. Πάλι ε, εγώ προσωπικά είμαι ο εισηγητής και πρόκειται για το μεταπηγημένο κρέας πουλερικών μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας αλλά και Ταϊλάνδης. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώνει τώρα. Εγκρίνεται λοιπόν ομοφόνος. Όλοι συμφωνείτε λοιπόν με την συμφωνία για το κρέας των πουλερικών. Όχι ότι εμένα μ' αρέσει, αλλά τι να κάνουμε, κάνει κανείς και θυσίες. Τώρα, ακολουθεί ο κανονισμός για κάτι που έχουμε ήδη ε, ψηφίσει, είναι το 18 για, την, ε, για, το, για το κοινό μάλλον δασμολόγιο. Πάλι εδώ είμαι εγώ ε, ο εισηγητής. Αρχίζει η ψηφοφορία εννοείται ηλεκτρονική. Τέλος. Πάλι ομόφωνη έγκριση. Και με μία αποχή. Uh, another Ας έρθουμε τώρα στα βαρέα βάρη που είναι το θέμα 19 έκθεση Καζάκ για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιαπωνίας. Και εδώ αρχίζω με την συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ωραία. Επαλήθευση λοιπόν για την 15. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τέλος. Και απεριφθιόνται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 Α, όχι. 26. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Ε, τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά Αποχές. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Πέρας. Και εγκρίθηκε. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο μαζί. 71 και 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14β υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 συμβαστική υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε καλύτερα. 93. Αρχίζει η ψήφος. Τέλος. Εγκρίθηκε εν τέλει. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92 υπέρ. Υπέρ, ε, κατά απόχέ Εγκρίνεται. Τώρα, οι λογική σκέψει. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ας επαληθεύσουμε την 5 δηλαδή ας την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά πέρας εγκρίθηκε και αυτή τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 7 κατά 7 λέει ο πρόεδρος Α, είναι παρόμοια, καλά 8 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η εννέα εκπίπτει έτσι δεν είναι. Δέκα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και έντεκα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψήφος επί όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει. Και τέλος. Και εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 3 αποχές Συγχαρητήρια στον κύριο Καζάκ για την επιτυχία της σημαντικής αυτής εκθέσεως. Τώρα. Το θέμα υπαριθμών 20 τροποποίηση παραρτημάτων, πρωτοκόλων Ευρωπαϊκή, ε, Συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κράτου του Ισραήλ. Υπάρχει μια τροπολογία, Πολ Μέρφυ, α την ψηφίσουμε, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο της γνωμοδοτήσεως. Συστάσεως μάλλον, συστάσεως. Πέρας. 25 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Το θέμα 21 Ωστόσο αποφασίσαμε χθε να κάνουμε ενδεικτική ψηφοφορία για να μπορέσει η ΑΦΕΤ να ψηφίσει. Εσείς και Λάιχτρη την εξηγήσετε τώρα γιατί. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε που διακόπτω την διαδικασία ψηφοφορίας, αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω ορισμένε ανακοινώσεις για το θέμα της ρήτρας προφύλαξης Safeguard. Προσήλθαμε στον τριμερή διάλογο την Δευτέρα με εκκρεμή διάφορα θέματα, τα οποία ωστόσο δεν διευθετήθηκαν ικανοποιητικά. Μένει ένα, μάλλον διευθετήθηκαν ικανοποιητικά. Υπάρχει ένα θέμα ακόμη, η κοινή δηλαδή η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου, Κομισιόν και δική μας και Κοινοβουλίου. Νομίζω βρισκόμαστε σε καλή πορεία για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Εξετάζεται προσεκτικά από την νομική μας υπηρεσία το ερώτημα. Θα υπάρξει και απόφαση του Συμβουλίου στο επίπεδο των μονίμων αντιπροσώπων στις 24 Δεκάτου. Και τότε μόνον θα καταστεί σαφές ποια θα είναι η τελική έκβαση. Άρα την τελική μας ψηφοφορία μπορούμε να την διεξαγάγουμε στις 6 Νοεμβρίου μαζί με Κολομβία και Περού. Και νομίζω ότι αυτό είναι και σκόπιμο. Θα ήθελα προσωπικά να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω τις και τους συναδέλφους που συνέβαλαν σημαντικά και ιδίως στον τριμηρή διάλογο όπου διατηρήσαμε τις θέσεις μας Ευχαριστώ βεβαίως και τη Γραμματεία και ιδίως τον επικεφαλής του γραφείου μου που πέρασε δύσκολες εβδομάδες. Ελπίζω ότι ωστόσο τώρα αυτά πέρασαν. Ο λόγος, και γι' αυτό θέλω να θέσω το θέμα αυτό, ο λόγος για τα προβλήματα αυτά είναι η παράξενη κατάσταση όπου 99,9% η συμφωνία είναι αρμοδιότητα της ίντα, ενώ η ΑΦΕΤ ορίζει το χρονοδιάγραμμα. Ε, πρέπει κάπως να δώσουμε μια λύση σε αυτό, ή θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ξανά στο μέλλον. Ευχαριστώ πάντω και πάλι. Οι διαπραγματεύσεις διεκδίκησαν καλώς, ήταν επιτυχής. Πρώτη φορά αφή έχουμε στα safeguards και κοινωνικά θέματα και αυτό είναι νέο για την Ευρώπη. έχουμε ένα είδος Κορέα συν. Ε, ευχαριστώ και για τη δυνατότητα να κάνω τις ανακοινώσεις αυτές και δεν πρόκειται βεβαίως να παρενοχλήσω περισσότερο την ψηφοφορία. Τουλάχιστον όχι τώρα. Παύλο, ναι, υποστηρίζω τα όσα είπε ο κύριος Λάιχτφριντ στο όνομα του Λαϊκού Κόμματος υποστηρίζουμε απολύτως τα επιχείρηματά του Ευχαριστούμε ιδιαίτερος τα μέλη της Γραμματείας για την εργασία τους των τελευταίων ημερών που πραγματικά ήταν πολύ εντατική για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε σήμερα και χάρη στην προσπάθειά τους αυτή μπορούμε όντως να ψηφίσουμε σήμερα. Αναμένω λοιπόν όσο το δυνατόν συντομότερα να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε και τα εκρεμή θέματα. Και ελπίζω ότι και τα άλλα δύο θεσμικά όργανα θα αποφασίσουν σύντομα. Ωραία. Είναι λοιπόν ξεκάθαρη κατάσταση. Έχουμε συμφωνήσει κάτι με την Κομισιόν, αλλά τώρα δεν συμφωνούμε με αυτό που συμφωνήσαμε. Κάπως έτσι βλέπω την κατάσταση. Άρα πρόκειται για ενδεικτική ψηφοφορία, άρα η οριστική ψηφοφορία θα γίνει αργότερα, τον Νοέμβριο. Μέχρι τότε Η Κομισιόν ελπίζω να καταβάλει τι απαραίτητε προσπάθειες για να ξεκαθαριστεί το περιεχόμενο της συμφωνίας. Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία αυτή. Τέλος. Εγκρίθηκε λοιπόν με 22 ψήφους υπέρ και 2 κατά. Συγχαρητήρια Κύριε Λάιχτφριντ. Μένει τώρα η γνωμοδότηση για την ΑΦΕΤ για ένα θέμα που είναι κατά 80% εμπορικό αλλά δεν είμαστε αρμόδιοι. Ο Παύλο Φάβα είναι εισηγητής. Υπάρχουν δύο τροπολογίες, η υπαριθμών 1 και η υπαριθμών 2 Αυτές είναι ταυτόσιμες και θα ψηφιστούν μαζί. Ας ψηφίσουμε λοιπόν τις δύο αυτέ τροπολογίες. Ψήφι υπέρ, κατά, απορρίπτονται. Τελική ψηφοφορία αρχίζει. Τέλος. Και όντως είμαστε υπέρ να δώσουμε τη συνένεσή μας δηλαδή στις συμφωνίες αυτές με 20 ψήφους υπέρ και 4 κατά. Τελειώσαμε με την ψηφοφορία και σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Οι εργασίες μας ωστόσο δεν τελείωσαν. Όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα, ας το πράξουν συντόμως. Και όσοι παραμένουν, να μπίνουν καθιστή. Well, when I say settle down, I mean settle down. Όταν, όταν λέω καθιστή, εννοώ καθιστή. hush, please. Joint items 23. Uh, Τα θέματα 23 και 24 τώρα σε κοινή συζήτηση. Ανταλλαγή απόψεων με τους ενδιαφερομένους για ένα παράλληλο θέμα. Εγώ είμαι εισηγητής και τα δύο. Παρακαλείστε όσοι κάνετε ουρά για να βγείτε έξω, να βγείτε έξω. This is about one of the many United Πρόκειται για θέμα Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, Committee for Europe, με συμμετοχή χώρων της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και άλλων για να βάλουν τα θεμέλια μιας οικονομικής συνεργασίας. Η Επιτροπή ε, Χερσαίων Μεταφορών της UNESCO για τη μεταφορά προσώπων και ε, εμπορευμάτων για χερσαίες μεταφορές δηλαδή υπάρχουν τρεις διεθνείς συμφωνίες των ΗΠΑ για τα μηχανοκίνητα οχήματα που διαχειρίζεται η UNESCO Στο πλαίσιο, γίνονται αντικείμενα διαχείριση στο πλαίσιο της UNESCO. Συζητούμε τώρα πρόταση της Κομισιόν με αντικείμενο την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφοφορίας κανονισμών της UNESCO των συμφωνιών του 1958 και 1998. Το σύστημα έγκρισης τύπων οχημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται όλο και περισσότερο στους κανονισμούς του UNESE που αντικαθιστούν την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, ταχύτερη έγκριση της νομοθεσίας θα επιτρέψει και ταχύτερη ανταπόκριση στις ε, κανονιστικές απαιτήσει. Το πλαίσιο της UNESE έχει θεμελιώδη σημασία για τη βιομηχανία μας και είναι και benchmark, ορόσημο, για τους κανονισμούς τους δικούς μας σε σχέση με συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και αποτελεί μια πολύτιμη βάση για ρυθμιστικές μετατροπές που είναι σημαντικές σήμερα όπου τα πιο σημαντικά κολλήματα στο εμπόριο δεν είναι πλέον δασμολογικά αλλά είναι κανονιστικές διαφορές. Και γι' αυτό νομίζω είναι επίκαιρη αυτή η ανταλλαγή απόψεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα την ανισχύσουμε ακούγοντας τον κύριο Ράμος Καρθία επικεφαλής του Vehicle Regulation για την εναρμόνιση των ε, κανονισμών σχετικά με τα μηχανοκίνητα οχήματα της ΟΝΕΣΕΜ σας ευχαριστώ, είστε εδώ. Σας βλέπω εδώ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης που μας δίνετε την ευκαιρία να σας εξηγήσουμε πώς ετοιμάζουμε τις ρυθμίσεις για τα μηχανοκίνητα οχήματα. Η εισαγωγή μου έχει διάφορα τμήματα. Το ένα είναι η στόχη και η δομή για να σας πληροφορήσουμε όσον αφορά το World Forum, τις δραστηριότητε μας. Το άλλο είναι οι συμφωνίες 1958 και 1998. Και τέλος, πώς οι συμφωνίες αυτές μπορούν να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο. Είναι μεγάλη κανονικά η παρουσίασή μου, αλλά μου δώσατε 10 λεπτά, οπότε θα την περιορίσω κάπως και να ξέρετε ότι αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να την έχετε ολόκληρη. Αυτό είναι λίγο ιστορική αναδρομή από το 1949 στη συνέχεια το 52, μετά είχαμε τις συμφωνίες 58-97. Το 2011 τώρα έχουμε τις προδιαγραφές ε, ποιότητας της αγοράς όσον αφορά τα οχήματα και για τα καύσιμα όμως, γιατί βέβαια χωρίς καύσιμα δεν ε, μπορεί να ε, λειτουργήσει ένα όχημα. Να παράδειγμα κάποιων δραστηριοτήτων του World Forum. Τις βλέπετε εδώ. Περιορισμός ε, των εκπομπών, για παράδειγμα. Ξεκινήσαμε το 1988 που είχαμε τα οξύδια του ζώτου και το διοξίδιο του άνθρακα. Μετά προχωρήσαμε στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και βλέπετε ότι η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα είναι 20% αν συγκρίνουμε με το 1988 υδρογονάθρακες λιγότερο από 5% Τώρα να δούμε την δομή της Ομάδας Εργασίας 29. Όπως ε, είπε, είμαστε με τα ενωμένα Έθνη, βασιζόμαστε στην, ε, έχουμε τη βάση μας μάλλον στη Γενέβη, έχουμε την Επιτροπή για τις Μεταφορές στην Ενδοχώρα και έχουμε επίσης και δομές για την εναρμόνιση. Έχουμε τέσσερις δραστηριότητες ε, για την προστασία, την γενική προστασία και με τις ομάδες εργασίας οι οποίες είναι όλες μόνιμες το breaks, η ρήπανση, η χορύπανση και ασφάλεια. Οι ομάδες εργασίας αυτές συμπληρώνονται και από ένα διοικητικό σώμα και από εκτελεστικές και διοικητικές επιτροπές για κάθε μία από τις συμφωνίες με τα Ηνωμένα Έθνη. Επιπλέον, βλέπετε κάτω-κάτω στη σελίδα αυτή ότι υπάρχουν και άτυπε ομάδες. Αν δηλαδή ένα θέμα χρειάζεται κάτι παραπάνω από 29 ε, συνεδριάσεις ε, το χρόνο στην ε, Γενέβη για τις δραστηριότητε μας, όταν υπάρχουν ειδικά θέματα που απαιτούν περισσότερο χρόνο, τότε το World Forum δημιουργεί ειδικέ ομάδες εργασίας οι οποίες ασχολούνται και αφοσιώνονται σε ένα ειδικό θέμα με όλε αυτές τις επίσημες και άτυπες ομάδες εργασίας ε, σήμερα δεν υπάρχει καμιά φωλή ότι αυτή τη στιγμή κάποια συνεδρίαση γίνεται κάπου στον κόσμο με ένα από αυτά τα όργανα. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, εμείς ε, στη Γενέβη έχουμε τρεις συμφωνίες και θα επικεντρωθώ εδώ στις δύο πρώτες, μια που αυτές έχουν σχέση με την κατασκευή των οχημάτων. Είναι η 58 που έχει να κάνει με την εκ των προτέρων έγκριση και πρέπει να ληφθεί υπόψη για το εμπόριο. Έχουμε 50 συμβαλόμενα μέρη και έχουμε 129 κανονισμούς. Η συμφωνία του 89 επίσης ε, παίζει ρόλο εδώ. Έχουμε μέχρι τώρα 12 ε, κανονισμούς από τα Ηνωμένα Έθνη. Οι συμφωνίες ε, πάντως ε, οι δύο αυτές να ξέρετε ότι έχουν πολλές διατάξεις που μοιάζουν. Γι' αυτό και μιλάμε για παράλληλη συμφωνία. Εδώ βλέπετε την, ε, πώς κατανέμονται οι συμφωνίες αυτές. Το πράσινο ανοιχτό είναι χώρες που μόνο συμμετέχουν στη συμφωνία του 1988 και στο κέντρο της Ευρώπης βλέπετε λίγο κίτρινο. Εκεί είναι χώρες που συμμετέχουν στη Συμφωνία του 50. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες μπίπτουν σε ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο που έχουν επίσης γίνει. Λέμε ότι είμαστε ένα σώμα ανοιχτό σε όλες τις χώρες των ΗΠΑ όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είδατε και στο χάρτη. Μη κυβερνητικέ και κυβερνητικέ οργανώσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Συμβουλευτικά όμως. Και οι αποφάσεις λαμβάνονται μόνο από τις κυβερνήσεις των συμβαλόμενων μερών. Υπάρχει και διαφάνεια στην οργάνωσή μας, γιατί όλα τα έγγραφα, ακόμα και εκείνα των άτυπων ομάδων εργασίας, ε, τα βρίσκει κανείς στην ιστοσελίδα μας. Θα επικεντρωθώ στις διατάξεις της Συμφωνίας του 58. Οι συμφωνίες των Ηνωμένων Εθνών προσαρτίζονται στις συμφωνίες των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα Σεβαλόμενα μέρη, και αυτό είναι σημαντικό εδώ, μπορούν να δεσμευτούν από όλους τους κανονισμούς ή από μερικούς από αυτούς. Όπως συνέβαινε και πριν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση ε, σε σχέση με την εθνική νομοθεσία. Μία νέα ρύθμιση υιοθετείται με τα δύο τρίτα των συμβαλόμενων μερών. Σας υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζει με 27 ψήφους δηλαδή όλων των χωρών μελών της. Μετά ξεκινάει η διαδικασία στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γενικός Γραμματέας κοινοποιεί ε, τις σχετικές ρυθμίσεις σε όλα τα μέρη και πρέπει να εφαρμόζονται στις χώρες αυτές, εκτός αν ε, για κάποιο λόγο υποβάλλουν κάποια αντίρρηση. Όλοι δεσμεύονται. Αλλά αν αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν κάποια ρύθμιση, πρέπει να το πούν. Σας ενημερώνω επιπλέον ότι πέρυσι εγκρίναμε πάνω από 130 τροποποίησεις στους 129 κανονισμούς που ήδη είχαμε. Οι ρυθμίσεις αυτές των Ηνωμένων Εθνών εφαρμόζονται χωρίς τροποποίηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορούν όλοι να τις αναγνωρίσουν συμπεριλαμβάνουν απαιτήσει επιδόσεων και προϋποθέσεις για την αμοιβαία αναγνώριση. Όλα τα οχήματα ε, περνάνε από τον έλεγχο αυτών. Υπάρχουν και άλλες χώρες όμως που εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις αυτές και που είναι στη διαδικασία να προσχωρήσουν στη συμφωνία. Τώρα θα σας μιλήσω για τη συμφωνία του 1988. Δημιουργήθηκε 1998. Δημιουργήθηκε από την άλλη μεριά του Ατλαντικού επειδή αποφάσισε να μην δεχτεί την αμοιβή αναγνώριση της συμφωνίας του 58. Η ιδέα όμως της συμφωνίας αυτής είναι ε, βασικά να έχει τις ίδιες διατάξεις, θα έλεγα τουλάχιστον κατά 90% με την συμφωνία του 58, αλλά η συμφωνία αυτή δεν έχει διοικητικές διατάξεις. Δεν ε, υπάρχουν ε, συστήματα έγκρισης. Μπορούν να παραχθούν δηλαδή οχήματα βάσει της συμφωνίας αυτής του 1998. Με τη συμφωνία του 1958 έπρεπε διοικητικά να εγκριθούν από όλες τις χώρες. Περιλαμβάνονται επίσης τεχνικές προδιαγραφές, μέθοδοι δοκιμής και επιδόσεις. Αλλά δεν υπάρχουν διοικητικές ε, προβλέψεις. Να τα συμβαλόμενα μέρη. Έχουμε μια δημοσίευση που μπορούμε να σας την μοιράσουμε. Αν επιθυμείτε δηλαδή να την έχετε, μπορούμε να σας την διαθέσουμε. Και θα ολοκληρώσω εξηγώντας σας πώς βλέπω και πώς οι ρυθμίσεις αυτές ε, του WP29 μπορούν να βοηθήσουν. Πρώτον υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή εάν εφαρμόσουν τις συμφωνίες αυτές οι χώρες μέλη υπάρχει πάντα κάποια ρύθμιση για όλα τα οχήματα. Έχουμε επίσης αποδείξει πόσο αποτελεσματικοί είμαστε για την προστασία. Θυμόσαστε τι σας είπα για τις εκπομπές ρηπογόνων ε, ουσιών. Πρόκειται βέβαια για μια δύσκολη και ακριβή δουλειά για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και εμείς στα συμβαλώμενα μέρη ε, προτείνουμε να αντικαταστήσουμε τις ε, όποιες δικές τους ρυθμίσεις που τους κοστίζει πολύ να τις ετοιμάσουν με τις δικές μας ρυθμίσεις που τους έχουμε σκεφτεί και αθετήσει. Οπότε κάνουμε συστάσεις. Πολλές φορές οι αναπτυσσόμενες οικονομίες λένε ότι οι δικές μας είναι υπερβολικά τεχνικές, είναι στο το επίπεδο, όμως μπορούν αν θέλουν να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ρυθμίσεις οι οποίες βρίσκονται σε ένα κατώτερο επίπεδο, που είναι δηλαδή προηγούμενες, πριν φτάσουμε τεχνολογικά σε τόσο, σε τέτοια σημεία χμής. Επίσης, οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται χωρίς τροποποίησης. Ενώ στην προηγούμενη συμφωνία μπορούσαν να υπάρχουν ε, τροποποίησεις. Σύμφωνα με τη συμφωνία του 78, εφόσον έχει εγκριθεί ένα όχημα σε μία χώρα α, πρέπει να εγκριθεί και στις υπόλοιπες οι οποίες, εγκρίνουν, οι έχουν προσχωρήσει στη συμφωνία αυτή. Δεν υπάρχουν διοικητικές διατάξεις, άρα ακολουθούμε τις διοικητικές διατάξεις των χωρών μελών. Με 2 τρίτα εγκρίνεται του 58, ενώ με συνένεση συμφωνία του 98. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για την έξοχη παρουσίαση. Έμαθα πολλά. Θα μελετήσω και τις διαφάνειές σας. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών έχουν εκπρόσωπο. Εδώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ καθηγητά για την παρουσίαση θα δώσω στον εμπειρογνώμονα να έρθει, που θα έρθει εκεί να κάνει την παρουσίαση, να πω μια λόγια πριν έρθει ο Άντολφ. Για τη βιομηχανία μας όταν γίνονται διαπραγματεύσεις για ελεύθερο εμπόριο, FTA, ε, ζητούμε να συμπεριλάβεται η συμφωνία του 58 στο παράρτημα. Πάντα το ζητάμε δεν θέλουν πολύ σημαντικά οι εταιρείε να το κάνουν, όπω η Ινδία, Μερκοσούρ, Κολομβία, κάποιε ΑΣΕΑΝ, χώρε ΑΣΕΑΝ, ο Καναδά και η Ιαπωνία σε κάποιο βαθμό. Εκεί με αυτού έχουμε προβλήματα και δυστυχώ έχουμε και πρόβλημα σήμερα με την εφαρμογή τη συμβάσεω αυτή τη συμφωνία με την Κορέα. Όλα αυτά είναι ευχολόγιο. Ελπίζουμε τελικά όμω όλα αυτά να πραγματοποιηθούν. Ο Ντόλφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ που με επιτρέπετε να αναφερθώ στη σημασία που έχει αυτή η συμφωνία και το πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Ντόφ Λάμπριξ είμαι, είμαι τεχνικός διευθυντής στην ACA. Εκπροσωπώ την ACA που είναι βασικός φορέας αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. 18 διεθνείς εταιρείες εκπροσωπούμε. Βλέπετε τις εταιρείε από κάτω στη διαφάνεια που εκπροσωπούμε. Έχουμε μεγάλο τζίρο. Παράγουμε πολλά. 427 δις σε φορολογικά έσοδα δημιουργήσαμε τα κράτη-μέλη. Σκοπός της σύντομης παρουσιάσεώς μου. Να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών Συμφωνίας για την αυτοκινητοβιομηχανία και το εμπόριο. Η αυτοκινητοβιομηχανία κινείται τάχιστα προς παγκοσμιοποίηση όλα πηγαίνουν πολύ γρήγορα. Τα οχήματα που διατίθενται στην παγκόσμια αγορά πρέπει να ανταποκρίνονται στις ντόπιε απαιτήσει των πελατών, αλλά πρέπει να υπάρχουν ε, τυποποίησεις της τεχνολογίας που απαιτείται και των προδιαγραφών. Η αυτοκινητοβιομηχανία συμμετέχει στην εναρμόνιση της νομοθεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά θέλουμε να καλύπτεται και ανάγκη του καινού ταυτόχρονα τα ωφέλη της εναρμονήσεως. φορά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Είναι σημαντικό, σημαντική εναρμόνιση για τους πελάτες. Θα έχουν αυξανόμενη επιλογή σε ανταγωνιστικές τιμές. Uh, για τις κυβερνήσεις χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα τους πόρους που διαθέτουν και είναι καλό και υποφελές για την προστασία των καταναλωτών διότι τυποποιημένη αυτή η νομοθεσία είναι η καλύτερη ρυθμιστική, αντιπροσωπεύει την καλύτερη ρυθμιστική πρακτική. Όλοι θα ωφεληθούν λοιπόν από την εναρμόνιση. Παράδειγμα εναρμόνισης τη τελευταία 20 ετία Είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά παρελθόν όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωσης είχαν τη δική του νομοθεσία καθεμία για τα οχήματα. Το 1985 ετοιμάσαμε το σύστημα διαφόρων τύπων οχημάτων που ετέθησε ισχύ το 1992. Έκτοτε, ένα όχημα που εγκρίνεται σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορεί να διατεθεί στην αγορά όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών. Και αυτό ήταν πολύ υποφελές για την μηχανία και για τη διοίκηση ήταν υποφελές και για τον καταναλωτή. Όλα τα οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπρεπε να συμμορφώνονται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές. Λοιπόν, το σύστημα έγκρισης τύπων οχημάτων EC που βλέπετε εδώ έχει πάρα πολλά, 55 ξεχωριστά συστήματα εγκρίσεων. Και ένα όχημα που συμμορφώνεται με, τα 55, με τις 55 αυτές απαιτήσει, παίρνει πιστοποιητικό ECWVTA και εγκρίνεται για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργήσε καλά το σύστημα, ξεκίνησε εργασία το 85, εφαρμόστηκε το σύστημα το 92 για τα επιβατικά οχήματα και για τα εμπορικά οχήματα Φέτος τον Οκτώβριο θα εφαρμοστεί. Τώρα δηλαδή, όπου να είναι. Ο Σονούπο. Η ίδια προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν και στον υπόλοιπο κόσμο. Το 1996 η αυτοκινητομηχανία ενετόπισε ότι είναι σημαντική η παγκοσμιοποίηση και ο φορέας Ε, ήταν η ομάδα εργασίας, το ε, η ομάδα εργασίας 29 στη Γενέβη θα μας βοηθούσε σαν φορέας. Και μετά τη συμφωνία του 58 επεξεργάστηκε η συμφωνία του 98 για να μπορέσει να, και, να συμμετάσχουν και ΙΠΑ. Είναι πραγματικά παγκόσμια επιτροπή. Το είδαμε αυτό το 2000 όπου η ονομασία Ομάδα Εργασίας 29 έγινε Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εναρμόνιση Νομοθεσίας για τα Οχήματα. Άλλαξε ο τίτλος. Και όπως είπε και ο προλαλής σας, η UNEC ε, χειρίζεται περίπου 130 ξεχωριστά νομοθετήματα για διάφορα συστήματα. Εσείς αναφέρετε 129. Ένα από τα 129. Αν κάθε χώρα επιλέξει για τα οχήματά της τεχνικές απαιτήσει εκτός του πλαισίου αυτού, μάλλον εάν ενταχθεί σε αυτό το πλαίσιο κάθε χώρα, πάμε στην παγκοσμιοποίηση ηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντικατέστησε τις διάφορες ξεχωριστέ οδηγίες η Ευρωπαϊκή Ένωση, διάφορου τύπου τύπους οχημάτων, με αντίστοιχου κανονισμούς Ευρωπαϊκής ο ΙΕ. Ε, και παροτρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσης να προσχωρήσει η φωνία του 58 και του 98, ούτως ώστε να υλοποιηθεί η παγκόσμια αρμόνιση. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει στόχο να παροτρύνουμε τι αρχέ να μην αναπτύσσουν η κάθε μία την δική της νομοθεσία. Όταν θέλουν να θεσπίσουν νέα νομοθεσία, θα πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή και να συζητείτε στο, στην ομάδα εργασίας 29 και να καταλήγουν σε παγκοσμίως αποδεκτές προδιαγραφές. Παράδειγμα, οι συζητήσεις οίκων στις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ταυτόχρονα η Ρωσία θέλει να κάνει αντίστοιχο σύστημα και λέμε στη Ρωσία, ξεκινήσει συζητήσει στην ομάδα εργασία 29 για να καταλήξετε σε παγκόσμια εμβέλεια νομοθεσία και οδηγία περί ανακυκλωσιμότητα. Θεσπίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα όλε οι χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, προσπαθούν να καταρτήσουν δικέ του απαιτήσει ανακυκλωσιμότητα και λέμε μην το κάνετε αυτό. Ας πάρουμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για ανακυκλωσιμότητα, να τη θέσουμε, να την υποβάλουμε στη Γενέβη και θα σπιστεί σαν κάτι παγκόσμιο. Να συμμορφώνονται τα οχήματα σε παγκόσμιο επίπεδο με τις διαγραφές, μειώνεται το κόστος έτσι, να υποφελείς τον καταναλωτή για τις κυβερνήσεις και θα είναι και πιο αυστηρές οι προδιαγραφές. Αυτά είχα να σας πω επί του θέματος και σας ευχαριστώ. Πράγματι, σας ευχαριστώ για αυτά που μας είπατε. Ας ξεκινήσει η συζήτηση. Ζητάει κανείς τον λόγο. Daniel Κάσπαρι, you are the Και Κάσπαρη, είστε σκιώδης, Λάγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία πράγματα κάπως με απασχολούν και ίσως ο Γενικός Γραμματεύς της ομάδας 29 μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις αφενός βρίσκω σωστό να έχουμε όσο δυνατόν παγκόσμιες προδιαγραφές ώστε να επιτυγχάνουμε και οικονομίες κλίμακος και να μην αναπτύσσονται κολλήματα στο εμπόριο μέσω των προδιαγραφών. Ο βέβαια είναι και πολύ ευαίσθητο το θέμα και κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να ρυθμιστεί, να ρυθμιστεί μοναχά με παρεμβάσει τη εκτελεστική εξουσία. Όταν πρόκειται για παράδειγμα για τον θόρυβο ή τα καυσαέρια, τότε βέβαια θίγονται και τα συμφέροντα των πολιτών. Και δεν έχω τόση εμπιστοσύνη σε εκπροσώπους των εκτελεστικών εξουσιών που διαπραγματεύονται στη Γενέβη και τα συζητούν μεταξύ τους δείξατε στην αρχή ένα πίνακα μείωση των εκπομπών καυσαερίων και τι έχει επιτευχθεί. Αυτά όμως δεν έγιναν οικειοθελώς μετά από ανάληψη δράσης της εκτελεστικής ουσίας στη Γενέβη. Τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέφεραν τις βελτιώσεις αυτές. Άρα το ερώτημα είναι πώς μπορεί να εξασφαλιστεί ώστε στο δρόμο προς μια εμβάθυνση σε μια εναρμόνιση, κάτι που είναι απαραίτητο, ταυτόχρονα να μην πάει χέρι με χέρι με μια αποδημοκρατικοποίηση. Πώς να διατηρηθεί δηλαδή η ανάμειξη και η συμβολή των κοινοβουλίων. Δεύτερο, υπάρχουν μεγάλοι εμπορικοί εταίροι, οι οποίοι παρόλο που είναι εταίροι στις διαπραγματεύσεις, στην ομάδα των 29, δεν θεωρούν ότι είναι σε θέση οι ίδιοι να αναλάβουν τους θεμελιώδεις αυτούς κανόνες, δηλαδή να υιοθετήσουν θεμελιώδεις αυτούς κανόνες. Έχουμε, για παράδειγμα, ψήφισμα, σήμερα το ψηφίσαμε για τη σχέση μας με την Ιαπωνία και αυτό είναι κρίσιμο. Το ότι η Ιαπωνία δηλαδή επίσης να δεχθεί τους εκκρεμούντες ακόμη κανονισμούς που είναι άνω των 100 για να έχει πρόσβαση στην αγορά. Πώς βλέπετε τις προοπτικές αυτές η Ιαπωνία δηλαδή στο προσεχές μέλλον να ανταποκριθεί στις απαιτήσει αυτές. Νομίζω, όπως είπα, ότι εκκρεμούν ακόμη 100 κανονισμοί και να τους υπογράψει. Υπάρχει έξτρα πίεση που ασκείται στην Ιαπωνία προς αυτή την κατεύθυνση. Τρίτο, πολλά εξαρτώνται από το ότι οι κοινέ προδιαγραφές πρέπει να προέλθουν, να προκύψουν από ένα κοινό κύκλο δοκιμασιών για φορτηγά αυτοκίνητα, αυτοκίνητα ή και μοτοσυκλέτες, για τον θόρυβο, για τις εκπομπές καυσαερίων, διοξιδίου του άνθρακος κλπ. Τι γίνεται εδώ. Δηλαδή, πότε θα έχουμε στα χέρια μας ένα κοινό κύκλο δοκιμασιών που να έχει εγκριθεί και να γίνεται δεκτό και από τις ΗΠΑ και από την Ιαπωνία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Επιθυμεί κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Από όσο βλέπω όχι. Α ακούσουμε την Κομισιόν τότε. Ποιο είναι, ποια είναι παρούσα, η κυρία Μαργαρίτα Τέρμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ομπλικάδα θεωρεί ότι οι δύο προτάσεις αυτές ε, είναι πολύ σημαντικές. Συμφωνούμε με τους ε, ενδιαφερομένους ότι η αποφάση που ελήφθησαν στα πλαίσια της ομάδας 29 στις οποίες ενεπλάκη και συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ σημαντικές στην προσπάθεια να πετύχουμε μια εναρμόνιση σε παγκόσμιο επίπεδο και εφόσον τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε όλο και περισσότερο να συμπεριλαμβάνουμε τους κανόνες τους διεθνείς και του ΟΗΑ και στην έγκριση τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σχετικό σύστημα το όλο θέμα γίνεται όλο και πιο σημαντικό και το σύστημα ε, των ψηφοφοριών του ε, θα πρέπει να εφηγραμμιστεί με την ε, συνθήκη της Λισαβόνα. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η παγκοσμιοποίηση χρειάζεται και παγκόσμιες προδιαγραφές. Ήδη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ολοκλήρωσή της ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια αγορά αν δεν έχουμε και νέες προδιαγραφές η εσωτερική αγορά αντικαθιστά εθνικές διατάξεις από ευρωπαϊκές διατάξεις. Άμα θέλουμε παγκόσμιο εμπόριο πρέπει να αντικαταστήσουμε προφανώς και τις εθνικές διατάξεις και τις ευρωπαϊκές διατάξεις από άλλες διεθνείς διατάξεις. Η πλατφόρμα λοιπόν είναι μια πολύ καλή ιδέα. Βέβαια, πρέπει να προσέχουμε πολιτικάνουμε. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ομοσπονδιακού τύπου που εγκρίνεται από τα δύο νομοθετικά σώματα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο διατηρεί το ρόλο του εγκρίνοντας ε, και αυτό και φέροντας νέες ιδέες για τις προδιαγραφές που εγκρίνονται. Νομίζω ότι ο Λάγκε ακριβώς πρότεινε ότι οι συμφωνίες διημερούς εμπορίου αποτελούν ε, έναν πάρα πολύ καλό μοχλό που μας επιτρέπει εντός εισαγωγικών να επιβάλλουμε Μπορεί το επιβάλλουμε να ακούγεται πολύ δυνατό, αλλά είναι για να πιέζουμε τους εμπορικούς μας ε, εταίρους να υιοθετούν τις προδιαγραφές αυτές. Έχουμε πιέσει πάρα πολύ την Ιαπωνία, για παράδειγμα, το ξέρετε. Είμαι συγγητής, οπότε ξέρω για τι πράγμα μιλάω. Και νομίζω ότι όλοι και οι Ιάπωνες γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία χωρίς ε, οι Ιάπωνες να δεσμευτούν να εγκρίνουν τη συμφωνία αυτικάς. Διότι ένα μεγάλο μέρος είναι οι διατάξεις για τα ευρωπαϊκά οχήματα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους, ε, μάλλον δεν υπάρχουν αρκετά που να κυκλοφορούν στην Ιαπωνία και δεν είναι δεν το θέμα των δασμών. Αν λοιπόν η Ιαπωνία δεχτεί ε, δεχτεί μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Και για τις Ηνωμένες Πολιτείες ισχύει κάτι αντίστοιχο. Γιατί υπάρχουν ε, διαφωνίες και όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο των οχημάτων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Είναι ένα στοιχείο κλειδί πάντως αυτό, πολιτικά και οικονομικά πολύ σημαντικό. Οπότε σας ευχαριστώ όλους για τη συνεισφορά σας στη συζήτηση αυτή. Και τώρα, μάλλον αργότερα, θα έρθω στο δικό μου σχέδιο έκθεσης για να αποφασίσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Τώρα, Ναι, ο κύριος Λάγκη έθεσε διάφορα ζητήματα και εγώ έκανα κάποια σχόλια. Οπότε, μήπως οι προσκεκλημένοι μας, οι τόσο εξέχοντες, θα μπορούσαν να μας ε, εκφράσουν την άποψή τους για τα όσα ακούστηκαν. Ο κύριος Ράμος, για παράδειγμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω ουσιαστικά τίποτα όσον αφορά τις ερωτήσεις στο αξιότιμο ευρωβουλευτή από την Γερμανία. Θέλω όμως να διευκρινίσω ότι το WP29 δεν ετοιμάζει ε, διατάξεις. Μην τον μπερδεύετε με την ε, Επιτροπή που ασχολείται με την Ευρώπη. Οι δικές μας οι διατάξεις εφαρμόζονται παγκοσμίως και γι' αυτό τις ονομάζουμε των Ηνωμένων Εθνών. Και ένας από τους στόχους της νέας τροποποίησης για τη Συμφωνία 58 είναι να λέει ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις χώρες ε, των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα για την τρίτη σας ερώτηση, αν μπορούμε να έχουμε ένα κοινό κύκλο για τις ε, εκπομπές των βαρέων, των ε, ε μοτοσακών υπάρχει δουλεύουμε πάνω σε ένα σχήμα που περιλαμβάνει και τον έλεγχο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δηλαδή πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο γιατί προσπαθούμε να συνδυάσουμε τις, ε, ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα για τα διάφορα οχήματα. Υπάρχει η Ιαπωνία, η Κίνα, ολόκληρη η Ευρώπη και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί μια συμφωνία. Πάντως προχωράμε. Η Ιαπωνία είναι συμβαλόμενο μέρος στη συμφωνία του 58 και σε εκείνη του 98 και σε θελοντική βάση εφαρμόζει τις Όταν όμω ε, η Ιαπωνία υιοθετεί μια από τι δικέ μα διατάξει, όλη η εθνική νομοθεσία ακυρώνεται και εφαρμόζεται τότε μόνο η δικιά μας. Είναι όπω όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση που πήρε μια απόφαση για το ΚΑΣ 51 που αντικαθιστά τις διάφορες οδηγίες με την ε, συμφωνία αυτή σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Παρακαλώ. Θα προσπαθήσω και εγώ να δώσω κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Μία από την απάντηση την έδωσε ήδη ο κύριος Ράμος. Ότι κάνουμε δοκιμές ε, για τις διάφορες δραστηριότητες σε εναρμονισμένο επίπεδο. Αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα για την ηχορύπανση. Σε ορισμένα σημεία της νομοθεσίας, τα συμβαλόμενα μέρη λένε ότι αυτό δεν πρέπει να το αποφασίζει η Γενέβη, είναι θέμα κυριαρχίας. Υπάρχουν ε, όμως δοκιμές που είναι εγκριμένες διεθνώς για την ηχορύπανση, αλλά τα επίπεδα αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο, γιατί δεν θέλουν να αποφασιστούν ε, στη Γενέβη. Έτσι λοιπόν η δοκιμή είναι ε, εναρμονισμένη, αλλά οι τιμές όχι. Το άλλο και γι' αυτό υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης πολλές φορές απέναντι στη Γενέβη σε σχέση με το κατά πόσο είναι καλή για όλους η νομοθεσία που αυτοί ετοιμάζουν. Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα προβλήματα από την αυτοκινητοβιομηχανία είναι ότι όταν ξεκινάς με παγκόσμιες ρυθμίσεις ε, είναι πολύ αυστηρές και κανένας δεν θέλει να παραιτηθεί από αυτό που έχει ο ίδιος για τον εαυτό του. Εμείς προσπαθούμε να είμαστε λογικοί. Τα συμβαλόμενα μέρη στην Γενέβη ε, εκπροσωπούν βέβαια τις χώρες τους και εννοείται ότι εκπροσωπούν και όπως λένε τα συμφέροντα των πολιτών τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ τους προσκεκλημένους μας για την παρουσία τους εδώ και για τόσα μας είπαν. Πάμε στο σημείο 24α τελευταίο σημείο έχει να κάνει με την ε, προσωρινή συμφωνία όσον αφορά αφρικανικές ε, χώρες ε, ανατολικές και νότου. Η προσωρινή συμφωνία, όπως ίσως γνωρίζετε, μεταξύ Μαυρικίου, Σεχελών, Μαδαγασκάρης και Ζιμπάμπουε υπογράφηκε και άρχισε να ισχύει στις 14 Μαΐου που μας πέρασε. Πρέπει να δώσουμε σύμφωνη γνώμη ακόμα. Είναι όμως ένα καλό νέο ότι η συμφωνία αυτή υπάρχει. Ο κύριος Κάσπαρη θα μας παρουσιάσει πάντως το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Επιτέλους ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Όλοι παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις των ΕΠΑ και Interim ΕΠΑ εδώ και πολλά χρόνια και καμιά φορά με δυσαρέσκεια βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι αντίθετη με τις ε, διατάξεις του καταστατικού του ΠΟΕ Από το 2002 έχουμε αναλάβει τις διαπραγματεύσεις για τα νέα Economic Partnership Agreements και το αργότερο από το 2008 χάσαμε και την τελευταία ευκαιρία, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, να επιτύχουμε μια πραγματικά νόμιμη κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, αυτό είναι και η δική μου αυτοκριτική, δεν έχουμε παρακολουθήσει τις προσπάθειες αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο να της δώσουμε κίνητρα, όθηση να δραστηριοποιηθεί περισσότερο. Πάντως υπάρχει τώρα μια συμφωνία ΕΠΑ με τις χώρες της Ανατολικής και με συμβρινής Αφρικής και νομίζω ότι πρέπει να καταβάλει προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει στη ρύθμιση της καταστάσεως αυτής, να συναχθούν δηλαδή ενδιάμεσες συμφωνίες και γι' αυτό παρακάλεσα να απελευθεί το θέμα αυτό στην σημερινή μερίσια διάταξη και χαίρομαι που είναι παρόντες και διάφοροι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων χωρών από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, Πιστεύω γνωρίζουμε ότι οι συμφωνίες αυτές εταιρική σχέσης δεν αποδίδουν πολλά για μας. Ωστόσο βοηθούν στην οικονομική ανάπτυξη των συμβαλωμένων με εμά χωρών. Αυτέ είναι που θα ωφεληθούν από την συμφωνία αυτή και γι' αυτό πολύ θα ήθελα τώρα να ακούσω τι απόψει των εκπροσώπων του. Ευχαριστώ. Όντως και εγώ νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να συζητηθεί το θέμα. Ας ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν πριν δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους. Ο Πίτερ Τόμσον. Καλημέρα Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που μου δίνετε να σας μιλήσω και ιδιαίτερος ευχαριστώ τον κύριο Κασπάρη, τον εξηγητή και για τα ανθαρρυντικά του λόγια για την επιταχυμένη αυτή διαδικασία. Θα ήταν ευπρόσδεκτο κάτι τέτοιο. Τον ευχαριστώ για τη δουλειά του. Έγινε αυτή σε πρώτερη φάση όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε αυτό το εγγραφό επισήμω. Όμως επεξεργάστηκε επ' αυτής της βάσης και εξεπώνησε τον Μάρτιο του 2009 ψήφισμα και ξέρω ότι εκείνο ηγήθηκε τη όλη προσπάθεια. Για τα έπα συμφωνεί, ε, Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε μια γενική συμφωνία, πλήρη συμφωνία για περιφερειακή ε, συμφωνία και με, το, και με την Παππούα Νέα Γουινέα στον Ειρηνικό αλλά αυτή η συγκεκριμένη συμφωνία είναι η πρώτη η οποία εφαρμόζεται προσωρινά στην Αφρική και γι' αυτό το λόγο προφανώς είναι μια σημαντική στιγμή και ευπρόσδεκτη. Πιστεύω ότι η συμφωνία με την περιοχή αυτή θα βοηθήσει να είμαστε σε, ε, να έχουμε επιτυχία όπως και με τη συμφωνία με τον Ελληνικό και με, την, με το Κάρα Φόρουμ. Και ελπίζουμε να υποστηριχθεί αυτή η προσέγγιση και ελπίζουμε και οι χώρες να συμμορφωθούν με αυτά που ανέλαβαν να κάνουν. Πριν από αυτή τη συνεδρίαση και ελπίζω να έχει ο κόσμος να ρίξει μια ματιά στο έγγραφο, διανύμαμε ένα έγγραφο με στοιχεία που αφορά τη συμφωνία αυτή. Ε, δεν θα αναφερθώ εκτενώς αυτό, αναφέρεται στα αγαθά που έχουν ε, απελευθερωθεί και σε κάποια άλλα στοιχεία. Στα γρήγορα να πω κάποια πράγματα η περιοχή ανατολική ε, και Νότιας ε, Αφρικής είναι περίπλοκη ζώνη και πολιτικά και οικονομικά υπάρχουν πολλές διαφορές στις διάφορες περιοχές. Αρχικά υπογράψαμε με τις 6 από τις 11 χώρες περιοχής τη Συμφωνία. Αλλά το 2009 μόνο τέσσερι υπέγραψαν την τελική συμφωνία. Ήμουνα με τη Βαρόνη Άστον όταν υπέγραψαν αυτές οι τέσσερις χώρες το 2009. Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Σεϊχέλες και Ζιμπάμπου ήταν οι τέσσερις χώρες. Οι δύο χώρες που απεσύρθησαν από την όλη εξίσωση, η Ζάμπια ε, και οι Κομόρες, ε, πιθανότατα δεν επέλεξαν να υπογράψουν τότε λόγω πολιτικών αλλαγών. Αλλά ίσως να υπάρχουν και άλλες εξηγήσεις. Τι κάνει αυτή η συμφωνία, κατά την άποψή μου, σαν προσωρινή συμφωνία καταρχάς ε, βελτιώνει και δίνει ασφάλεια δικαίου και ευχαριστώ τον κύριο Κασπάρη που αναφέρθηκε στο τμήμα που αφορά τη συμμόρφωση του κανόνε ΠΟΕ. Λέγω, παρέχει ασφάλεια δικαίου για συνεχή πρόσβαση στην αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Και επ' αυτού βασίστηκε η εργασία πολλών εταίρων το 2007. Δημιουργεί εταιρική σχέση για την ανάπτυξη. Ε, σύμφωνα με την ευρύτερη διευθέτηση που έχουμε τις χώρες αυτές στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού, ε, εστιαζόμενη πάντα επί των εμπορικών θεμάτων, δίνει και άλλο ένα βήμα προς περιφερειακή ολοκλήρωση, εξορισμού, έχουμε υποσύνολο των χωρών, αλλά το γεγονός ότι πήραν συλλογικά αυτή την απόφαση, αυτό καθε αυτό, είναι μια ευπρόσδεκτη κίνηση. Και τέλος, παρέχεται επίσης εδώ και η βάση για βαθύτερη και ευρύτερη ελπίζουμε συνεργασία σε περίπτωση γενικής συμφωνίας, κάτι για το οποίο θα πρέπει να εργαστούμε. Στα πλαίσια της ε, υλοποίησης και εφαρμογή να επενθυμίσω ότι στο Μαυρίκιο το 2009 όταν υπογράφηκε συμφωνία έγινε μια διάσκεψη ε, ε, που μας βοήθησε να δούμε πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί η συμφωνία και φέτος επίσης, αρχές του έτους, ετοιμάσαμε σεμινάριο με θέμα την εφαρμογή της συμφωνίας. Έλαβε χώρα αυτό το σεμινάριο τον Μάρτιο και είχε εστιαστεί επί των επιχειρηματικών κύκλων των τεσσάρων χωρών. Αξίζει να πούμε ότι ελπίζουμε να διεξαχθεί ενακτήρια συνεδρία της Επιτροπής δηλαδή είναι ο φορέας που προβλέπεται τη συμφωνία τον επόμενο, την επόμενη εβδομάδα ε, ελπίζοντας ότι θα ρυθμιστούν κάποιες λεπτομέρειε και αμέσως μετά ελπίζουμε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε για τα αποτελέσματα της συμφωνίας στις 19 Οκτωβρίου. Να προσθέσω και κάτι τελικό, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρέασε την κατάσταση στις στάσεις που συμπεριλάβαμε στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2009 ε, έλαβαν υπόψη, ελήφθησαν υπόψη στις γενικές διαπραγματεύσεις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά και με τα χαρά να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις που θα έχετε σαν αποτέλεσμα της πρωινής συζητήσεως. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος αυτό το έντυπο με τα στοιχεία έχει διανεμηθεί πράγματι, περιέχει τα βασικά χαρακτηριστικά της προσωρινής συμφωνίας, τα αγαθά που απελευθερώνουν, τα αγαθά που εξαιρούνται και όλες αφορούν τις διαπραγματεύσεις και τα θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας. Σύντομο μεν, πλήρες δε το έγγραφο. Όπως τα γνωρίζετε, το επίπεδο απελευθέρωσης και χωρών που συμμετέχουν ε, το επίπεδο απελευθέρωσης ποικίλει ανάλογα με τις χώρες όπως στη Μαδασχάρη και στη Ζιμπάμπουε έχουμε 80% φιλελευθερωποίηση. Μαυρίκιος, Σεϊχέλες πάνω από 95%. Αυτό ταιριάζει και με την προσέγγιση μας όσον αφορά την ασύμετρη προσέγγιση. Ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των εταίρων μας στην Αφρική. Έχουμε και εκπροσώπους δύο χωρών. Είναι σύμπτωση. Είναι λιγότερο ανεπτυγμένες που εκπροσωπούνται Έχουμε τον πρεσβευτή της Ζιμπάμπουε, την πρέσβυρα της Ζιμπάμπουε μάλλον. Α, δεν κατέφθασα ακόμα. Είναι εδώ ο υπεύθυνο ε, εκπρόσωπος της Μαδαγασκάρης για εμπορικά θέματα. Α, δικό μου λάθος. Επιτετραμένο τη. Επιτετραμένο του Μαυρικίου ή επιτετραμένη. Η κυρία Σαμπρίνα Μούτου είναι εδώ μαζί μας. Ναι, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Θέλετε να πάρετε το λόγο μήπως. Ορίστε. Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ που μας καλέσατε να σας μιλήσουμε και να εκφράσουμε και τις απόψεις των χωρών μας όσον αφορά αυτή την Συμφωνία Οικονομικής ε, Συνεργασίας. Ευθύς εξ αρχής, ζητώ συγγνώμη από πλευρά του πρεσβευτού, δεν είναι εδώ, είναι σε αποστολή στο Μαυρίκιο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα είμαι σύντομη, διότι ήταν πολύ καλή σύνοψη που έκανε ο συγητής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο κ. ο συνάδελφος είναι εδώ, ο οποίος θα μιλήσει εάν τυχόν χρειαστούν κάποιες διευκρινήσεις αργότερα. Όπως υπόθηκε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέσσερις χώρες υπέγραψαν το Μάιο 2012 και επικύρωσαν τη συμφωνία και είναι μια πρωτιά αυτή στην Αφρικανική Ήπειρο θεωρείται ακρογωνίως λήθος για μια πλήρη συμφωνία, γενική συμφωνία. Όπως τα γνωρίζετε, ξεκίνησε η εφαρμογή, είναι κάτι πολύ καινούριο και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη δομή και τις διαδικασίες και τον, εσωτερικό κανονισμό της ε, Επιτροπής για την υλοποίηση συμφωνίας. Και περιμένουμε τη 19 του μηνός, την επόμενη εβδομάδα, να γίνει η ε, εναρκτήρια συνεδριασης της Βρυξέλλες. Η αντιπροσωπεία μου θα ήθελε να εκφράσει την εκτίμησή της όσον αφορά τον κανονισμό 1528 για την πρόσβαση στην αγορά, όπου εκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ε, εγκρίνει μια παράταση διετή. Αυτό θα δώσει μια ανάσα ε, στους διαπραγματευτές, κυρίως για τις χώρες που δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία. Θα αναφερθώ στις απόψεις του Μαυρικίου, όπως μου ζήτησε ο καθηγητής να σας πω. Ο Μαυρίκιος θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία είναι σημαντικότατη και περιμένουμε ότι θα είναι επωφελής και για τα... και τις δύο πλευρές υπό την προϋπόθεση ότι οι διαπραγματεύσεις θα λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες τις αναπτυξιακές ε, τις ιδιαιτερότητες των χωρών. Η συμφωνία είναι επίσης σημαντική για το Μαυρίκιο ε, διότι πιστεύουμε ότι με τη μεταρρύθμιση της συμφωνίας ε, έβγαινε εκτός των συμφωνίας γενικευμένων προτιμήσεων ο Μαυρίκιος και αυτή η συμφωνία θα είναι υποφελής όχι μόνο ε, για όλη τη χώρα ε, ε, αλλά και για τους εξαγωγείς του Μαυρικίου διότι θα έχουν ευρύτερη πρόσβαση για πολλά προϊόντα. Θα έχουν ευρύτερη πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να είναι αποτελεσματική συμφωνία και να έχει στόχο τον προσανατολισμό που είναι βασική προϋπόθεση της Συμφωνίας Κοτονού ο Μαυρίκιος πιστεύει ότι χρειάζεται να υπάρχει κατάλληλο περιβάλλον για απελευθέρωση του εμπορίου. Είναι σημαντικό αυτό και οι χώρες θα πρέπει να βοηθηθούν στις προσπάθειες που κάνουν για να ενταχθούν καλύτερα στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Όμω, με του νέου προσδιορισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το εμπόριο και τη χρηματοδότηση για το εμπόριο και την ανάπτυξη, θεωρείται σαν μικρή νησιωτική χώρα ο Μαυρίκιο και μια χώρα με μεσαία έσοδα και με αυτή την προσέγγιση ως τελικά να βρεθεί σε δυσχερή θέση ο Μαυρίκιος. Και αν αφαιρεθεί υποστήριξη για τη μετάβαση την οικονομική της χώρας μας σε αυτή τη φάση, αυτό θα υπονόμευε τις προσπάθειες που κάνουμε για ανάπτυξη και όσα έχουμε πετύχει στην προσπάθειά μας και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια οικονομική ε, ύφεση, ε, υπαναχώρηση. Και αυτό θα ήταν αντίθετο με τους στόχους αναπτυξιακού συμφωνίας Κοτονού και με την προσέγγιση της ε, Ευρωπαϊκής Ενώσης όσον αφορά τις διάφορες συμφωνίες που έχουν συναυθεί. Αυτή είναι η πρώτη συμφωνία, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αφρικανική Ήπειρο. Η αντιπροσωπεία μου πιστεύει ότι ίσως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα παράδειγμα, σαν ένα όχημα για να δημιουργηθούν και άλλα μορφώματα στην Αφρικανική Ήπειρο και να κινηθούμε προς μια πλήρη συμφωνία, γενική συμφωνία διότι υπήρχαν ανησυχίες και δισταγμοί να υπογράψουν τη συμφωνία αυτή ε, διάφορες χώρες για να γίνει αυτό αξιότιμα μέλη η συμφωνία πρέπει να γίνει ελκυστική για τους άλλους θα πρέπει να παρασχεθεί η αναγκαία βοήθεια του ώστε να προετοιμαστούν οι χώρες να επιφέρουν διαθετικές αλλαγές ε, να εφαρμόσουν εμπορικές πολιτικές και να βελτιώσουν τις υποδομές και την ανταγωνιστικότητά του ώστε να αρπάξουν τις εμπορικές ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο πιστεύουμε ότι είναι κρισίμου σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει και άλλους πόρους ούτως ώστε ε, να βοηθηθεί η εφαρμογή της συμφωνίας ε, και κυρίως ε, το κόστος προσαρμογής. Ο Μαυρίκιος θέλει να διαπραγματευτεί μια πλήρη συμφωνία, κάτι που το αποδείξαμε. Διότι ήδη υπογράψαμε, απελευθερώσαμε μάλλον 96% των δασμών μας. Αξιότιμα μέλη, Δράτω με τις ευκαιρίες να σας επιστήσω την προσοχή επί ενός θέματος που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες στο Μαυρίκιο. Αφορά την σόρευση προέλευσης πρώτων υλών που προέρχεται από χώρες εκτός ΕΟΚ. Σύμφωνα με τις συμφωνίες ΕΠΑΡ, οι, οι, οι χώρες που θέλουν χρειάζεται τελωνιακή συνεργασία για, για πρώτες ύλες που έρχονται από χώρες εκτός ΕΟΚ. Ε, αυτό είναι κάπως δύσκολο σε αυτή τη φάση, διότι οι περισσότερες από αυτές τις χώρες είτε δεν γνωρίζουν τη συμφωνία και τη διατάξη συμφωνίας, είτε δεν έχουν τις αναγκαίες δομές εντός των τελωνιακών τους ε, αρχών για να συναυθείτε τη συμφωνία. Είναι μια πρόκληση. Πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να εξασφαλίσουμε την πρόσβασή μας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι καταβάλλονται, απαιτούνται προσπάθειες μάλλον στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως για τα επίμαχα ζητήματα. Εμείς παραμένουμε αισιόδοξοι ε, σαν χώρε και πιστεύουν θα βρεθεί λύση. Έχουμε έξοχες σχέσεις, ιστορικές έξοχες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε την πεποίθηση ότι Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιδείξει την αναγκαία ευελιξία, ούτως ώστε τελικά να έχουμε θετικά αποτελέσματα με στόχο την ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Έχει ήδη αφηχθεί και η πρέσβυρα της Ζιμπάμπουε, η κυρία Μουτσάδα. Καλώς ήλθατε και έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου προσφέρετε την ευκαιρία να συνδιαλεχθώ με την Επιτροπή σας Εξωτερικού Εμπορίου. Η χώρα μου παραμένει δεσμευμένη στην εφαρμογή της ε, συμφωνίας με την Ευρώπη και για την κύρωση της Interim ΕΠΑ, e διότι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στη βασισμένη συμφωνία του Κοτονού είναι και ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός. Από... Επειδή η συμφωνία αυτή είναι και η πρώτη στην Ήπειρό μας, θα αποτελέσει και ένα κίνητρο και για άλλες χώρες να προσέλθουν στι συμφωνίε αυτές, μαθαίνοντα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι σωστό το πρόγραμμα αυτό να αποδειχθεί επιτυχές ώστε να γίνει ευκαιστικό και για άλλες χώρες. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων χρειάστηκε χρόνο ώστε πολλά από τα ωφελήματα που αναμέναμε στην αρχή με την αναθεωρημένη συμφωνία Κοτονού έχει χρειαστεί να αναθεωρηθούν ορισμένες από τις εξελίξεις επέλασαν αρνητικά στα ωφελήματα που αναμέναμε από τη Συμφωνία. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει σοβαρά την εφαρμογή και προσαρμογή που είναι, απαραίτητες, που είναι απαραίτητα για τις συμφωνίες αυτές με τις χώρες ΕΣΑ, Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, ώστε οι, συμβαλόμενα μέρη να μπορέσουν να προσαρμόσουν τις υποδομές τους στις παραγωγικές τους ικανότητες. Οι προσπάθειες που κάνουν οι συμβαλόμενες χώρες δείχνουν και την δέσμευσή τους για να προχωρήσει η διαδικασία και χρειάζεται βεβαίως ευκαμψία και επιθυμία προσαρμογής και από τις δύο πλευρές. Όταν συζητήθηκαν πρώτη φορά οι συμφωνίες ΕΠΑ, τώρα μάλλον στην, ε, την προτεραία της εφαρμογής δεν υπάρχει καμία δέσμευση για το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τουλάχιστον έχει γίνει δεκτό ότι έχουμε μια επιτροπή ανάπτυξης που εξετάζει τα θέματα αυτά. Οι προκλήσει που αντιμετωπίζουμε έχουν ω εξή. Η έλλειψη δεσμευτική συμφωνίας γίνεται αντιληπτή από τις χώρες ΕΣΑ διότι χρειάζονται συγκεκριμένες προσβάσεις σε πόρους για να προωθηθεί η ανάπτυξη, η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη. Η, τα συμβαλόμενα μέρη της ΕΣΑ σημειώνουν με ανησυχία πόσο αργά προχωρούν οι διαπραγματεύσεις και επίσης την έλλειψη επιθυμίας από πλευρά των συμβαλωμένων μερών για την εφαρμογή ορισμένων ιδιών που είχαμε ε, θεωρήσει ότι θα περιληφθούν στις ε, ΕΠΑ. Εμείς παρακαλούμε να αναλάβετε πλήρη, πλήρη την ευθύνη των υποχρεών σας για να εφαρμοστούν οι συμφωνίες. Γνωρίζουμε και ποιες αλλαγές προέκυψαν μετά από την συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Για παράδειγμα, στην κοινή αγροτική πολιτική, που για τη δική μου χώρα, που είναι αγροτική χώρα, σημαίνει σημαντικούς περιορισμούς η Ζιμπάμπουε θα χρειαστεί πόρους για να αναπτύξει βιομηχανίες της. Έχουμε ήδη υποστεί κυρώσεις δεκαετίας. Χρειαζόμαστε λοιπόν πόρους για να εξασφαλίσουμε προστιθέμενη αξία, να στερεώσουμε την εξαγωγική μας ικανότητα, διότι οι συμφωνίες αυτές αποτελούν αμφίδρομο. Χρειάζεται μάλλον η μείωση των επενδύσεων έχει επιβαρύνει την τοπική βιομηχανία. Και έτσι καθυστερούμε απέναντι στις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Και αυτό μειώνει την παραγωγικότητα των ε, τοπικών βιομηχανιών. Πιο συγκεκριμένα, η Ζιμπάμπουε χρειάζεται τεχνολογική υποστήριξη για να εξασφαλίσει την απαραίτητη υποδομή, να μπορέσει να αναπτύξει τις δυνατότητές της. Η υποστήριξη ΕΠΑ πρέπει να προσφέρει τεχνολογική υποστήριξη στους τομείς εκείνους που έχουμε οριοθετήσει για να αυξηθεί και η αποδοτικότητα. Κύριε Πρόεδρε, μετά από την αναστολή της εφαρμογής του άρθρου 96 η Ζιμπάμπουε είχε ελπίσει ότι η δράση αυτή θα επέτρεπε στην χώρα να μπορέσει να εμπορευτεί πιο ελεύθερα. Όμως εξακολουθούν και υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, για παράδειγμα για την πώληση αδαμάντων, καθώς και άλλοι περιορισμοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υπαναχωρεί από τις ε, δεσμεύσεις της. Άλλος τομέας που μας εκπλήσει είναι η εντύπωση που έχουμε για τις πολιτικοποιημένες αποφάσεις της διαδικασίας Κίμπερλε που περιορίζουν σημαντικά την πώληση διαμαδιών από τη Ζιμπάμπουε. Ενώ ήδη η Υπουργική Διάσκεψη του Μαΐου έχει ζητήσει την κατάργηση όλων των κολλημάτων και περιλαμβάνεται μάλιστα και στο σημερινό τύπο της Ζιμπάμπουε, όπου ο Πρωθυπουργό προβαίνει σε σχετική δήλωση. Και η Επιτροπή σας που είναι σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εμπορίου, να δείξει ευαισθησία στα θέματα αυτά, τα οποία εξακολουθούν να υπονομεύουν την ανάπτυξη της χώρας μας. Ενώ προβλέπεται συνεργασία και στη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ζιμπάμπουε αποτελεί και μέρος των περιφερειακών συνασπισμών της Μεσημβρινής Αφρικής με στόχο τη φιλελευθερωποίηση ώστε να φτάσουμε σε μια τελωνιακή ένωση. Ενώ μέχρι τώρα η εξέλιξη έχει επιβαρύνει μια ήδη εύθραυστη βιομηχανία. Εμείς με τις ενδιάμεσες συμφωνίες προβλέπουμε και ελπίζουμε σε αυξημένο εμπόριο μεταξύ Ζιμπάμπου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ αυτό που βλέπουμε τώρα είναι στρεβλώσει του ανταγωνισμού, αν δεν μπορέσουμε να επανεξοπλίσουμε τη βιομηχανία μας. Βλέπουμε λοιπόν ανάγκη για κάποια μέτρα θεραπευτικά των στρεβλώσεων. Συνεπώς, ο ιδιωτικός τομέας μαζί με το γενικό δημόσιο τομέα ζητούν την εφαρμογή μέτρων κατά του ντάμπινγκ και των επιδοτήσεων των εξαγωγών που έχουν βλάψει την βιομηχανία τροφίμων μας, για παράδειγμα. Αυτά συνοπτικά. Οι ανάγκες μας πρέπει να βασιστούν σε ενισχυμένη ανάλυση των δασμολογίων. Υπάρχει χώρος για την αναθεώρηση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Χρειάζεται, όπως είπα, και τεχνική υποστήριξη. Πάλι εδώ θεωρούμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να αρχίσουμε τη διαδικασία ελευθέρωσης. Αλλά βεβαίως χέρι με χέρι με κάποια εργαστήρια ευαισθητοποίησης που θα συμμετέχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, αλλά και για την πλήρη κατανόηση των κανονισμών που δεσμεύουν τις ε, σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Εμπορική Αρχή της Ζιμπάμπουε και το αρμόδιο Υπουργείο και η Βιομηχανία. Καθώς και άλλοι θεσμοί όπως η Επιτροπή Δασμών και Ανταγωνισμού, η Υπηρεσία Στατιστικής και άλλα όργανα και οργανισμοί που ασχολούνται με εμπορικά ε, θέματα, όπως και ο ΠΟΕ. Επίσης, απαραίτητα για μας είναι η εκπαίδευση στα συστήματα αυτά. Καθώς βέβαια και με συμμετοχή του οργανισμού τυποποίησης στη Ζιμπάμπου, έτσι ώστε να εφαρμοστούν και τα απαραίτητα φυτογειονομικά μέτρα που προκύπτουν και από τις περιφερειακές πολυμερείς συμφωνίες μας καθώς και από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. θέλαμε να δούμε ενίσχυση της εκπαίδευσης για την εφαρμογή των προδιαγραφών ποιότητας καθώς και checkpoints στα σύνορα. Τεχνολογική υποστήριξη που να μας επιτρέψει να ενισχύσουμε την υποδομή μας και να επιτύχουμε τη διασύνδεση μεταξύ μικρών μεσαίων και μεγάλων βιομηχανιών. Ως χώρα αν παραμένουμε δεσμευμένοι στη συνέχιση των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και μέσα στα πλαίσια της ομάδας ΕΣΑ για να εφαρμοστούν πλήρως οι συμφωνίες ΕΠΑ και νομίζουμε ότι τότε πια θα αναπτυχθούν πλήρως τα ωφελήματα που αναμένουμε από τις συμφωνίες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Ο επιτετραμένος τώρα της Μαδαγασκάρης έχει το λόγο, ο κύριος Ιμπραήμ Νορμπέα Ρισάρ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ που μας προσκαλέσατε. Προκειμένου να σας μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό για τις οικονομίες μας. Θέλουμε να σας πούμε επίσης και δύο λόγια για την δικιά μας θέση απέναντι στο ζήτημα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό πράγματι γιατί η Μαδαγασκάρη είναι μεν μία χώρα λιγότερο ανεπτυγμένη και θα μπορούσε να είχε και άλλες επιλογές. Έχει συμφωνία εταιρική σχέσης οικονομικής ε, όμως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και σε Χέλες, ο Μαυρίκιος και η Ζιμπάμπουε. Για πολλούς λόγους. Καθαρά νομικά μιλώντας, ε, δεν μπορούμε να πάμε αντίθετα στο ρεύμα. Όλοι γνωρίζουν ότι η συμφωνία ΑΓΑΤ απαιτεί μια εξέλιξη όσον αφορά τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε λοιπόν να αποτελέσουμε εμείς εξαίρεση. Αυτό είναι προφανές. Οικονομικά μιλώντας, η Μαδαγασκάρη είναι πεπισμένη ότι η ενδιάμεση συμφωνία είναι μια συμφωνία από την οποία θα υποφεληθεί η οικονομία μας. Συνεπώς, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων των εταιρικών σχέσεων είτε των προσωρινών είτε μια πλήρου τέτοια συμφωνία εταιρική σχέση διέπεται από το πνεύμα αυτό ακριβώς. Η Μαδαγασκάρη πολλές φορές μέχρι τώρα έχει πει ότι δεσμεύεται να διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σχέδιο, μια συμφωνία προσωρινής οικονομικής εταιρικής σχέσης. Το 2007 μονογράφησε την διάμεση συμφωνία με το άνοιγμα το δασμολογικό για 15 χρόνια. Η προσχώρηση της Μαδαγασκάρης ε, ε, ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2009 με την τελική υπογραφή. Μετά την υπογραφή αυτή, οι αρχές στις 3 Ιουνίου του 2011 ενημέρωσαν το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Στις 8 Νοεμβρίου τέλος του 2011 οι αρχές της χώρας μας επιβεβαίωσαν ότι συμφωνούν για ε, κοινή κοινοποίηση στον ΠΟΕ. Για μας όμως η ενδιάμεση συμφωνία αποτελεί μόνο ένα σταθμό. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και να συνυπογράψουμε μια πλήρη συμφωνία κάποια μέρα. Γι' αυτό και είμαστε σε διαπραγματεύσεις για μια τέτοια πλήρη συμφωνία και στις διαπραγματεύσεις αυτές συμμετέχουμε ενεργά. Η Μαδαγασκάρη θέλει να καταλάβει, μάλλον θέλει να υπάρχει ένα τμήμα για την ανάπτυξη από το οποίο η ενδιαφερόμενη χώρα θα μπορεί να υποφεληθεί πλήρως. Πρόκειται για μια συμφωνία ισορροπημένη, δίχως άλλο. Μόνο αν είναι ισορροπημένη συμφωνία μπορούμε πραγματικά να αποφεληθούμε πλήρως από μια τέτοια συνολική ε, συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις διάμεσες συμφωνίες που έχουμε υπογράψει μέχρι τώρα, πιστεύουμε ότι τα οικονομικά συμφέροντα της ε, Μανταγασκάρης προστατεύονται. Παρόλο που θα υπήρχε κάποιο περιθώριο για βελτίωση, η συνάδελφος από το Μαυρίκιο το υπογράμμισε γιατί υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, υπάρχουν κάποια πραγματάκια για ορισμένες πτυχές στι συμφωνίε αυτές. Συνεπώς οι διατάξεις επιδέχονται βελτίωση. Αλλά λέω πάντως ότι τα συμφέροντά μας σε έναν βαθμό τουλάχιστον προστατεύονται. Η μείωση των ε, δασμών έχει να κάνει με τη μείωση της τιμής των πρώτων υλών και με τον εξοπλισμό. Οι ευαίσθητοι τομεί έχουν αποκλειστεί από το χρονοδιάγραμμα μείωσης των τιμών για τη Μαδαγασκάρη. Συνεπώς, χοντρικά, τουλάχιστον να πως έχει η θέση της Μαδαγασκάρης όσον αφορά την διάμεση συμφωνία και όσον αφορά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη συμφωνία. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά για να τελειώσω θέλω να σας επιβεβαιώσω εδώ τη στήριξη της Μαδαγασκάρης σε όσα ακούσαμε και στις ανησυχίες των προλαλισσόντων. Διότι τελικά προκειμένου να πετύχουν οι συμφωνίες αυτές οι οικονομίες μας χρειάζονται στήριξη για να κάνουμε τις προσαρμογές εκείνες που χρειάζονται ώστε να επωφεληθούμε όσο γίνεται καλύτερα από τις συμφωνίες αυτές. Πρόκειται για συμφωνίες εταιρική σχέσης, έτσι. Ε, δεν είμαστε όμως στο ίδιο επίπεδο. Άρα χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις, κάποιες διορθώσεις από τη δικιά μας την πλευρά, ώστε να βρεθούμε αν όχι στο ίδιο επίπεδο με την ευρωπαϊκή πλευρά, αν μη τι άλλο να μπορούμε να επωφεληθούμε πλήρως από τις συμφωνίες αυτές. Συνεπώς, οι ανησυχίες που ακούσατε ισχύουν, είναι και δικές μας, τις ημεριζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Α, και η αντιπροσωπεία μου, εγώ ήρθα εδώ με κάποιους συναδέλφους που ασχολούνται άμεσα με τα θέματα αυτά και οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας αν έχετε ερωτήσεις να σας απαντήσουν. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ε, για τις ερωτήσεις τώρα. Ο Πολ Μέρφυ, πρώτα απ' όλα από την ΓΚΟΕ. Παρακαλώ, έχετε και το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για όλες τις παρουσιάσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα. Οι συζητήσεις αυτές για τις ενδιάμεσες συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές. Αξιολογούμε έτσι πώς έχουν τα πράγματα όσο προχωράει η διαδικασία. Και ακριβώς επειδή γίνονται κάπως κεντρικά από την Επιτροπή για την Αφρική, η πραγματικότητα μερικές φορές είναι ένας εκβιασμός για, προς τις χώρες αυτές, κατά πόσο δέχονται ή όχι τις διάμεσες συμφωνίες, αλλιώς ε, ακυρώνονται. Είναι ένα συνεχές στρες δηλαδή, που έχουν οι χώρες αυτές κάθε φορά που πρέπει να υπογράψουν νέες μεταβατικές συμφωνίες. Εγώ δεν συμφωνώ με τη θετική αξιολόγηση που από ό,τι φαίνεται αποτελεί και την ε, γενική αντίληψη στην αίθουσα ότι βοηθούν στην ανάπτυξη, στην περιφερειακή ολοκλήρωση κτλ. Ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα με τις συμφωνίες αυτές είναι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο ότι εξακολουθεί να υπάρχει ελεύθερο εμπόριο προς το συμφέρον των μεγάλων επιχειρήσεων που βέβαια ντύνονται με το μανδύα της προδευτικότητας. Είναι απίστευτο η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου να λέει ότι πρόκειται για επιτυχία όσον αφορά την ε, ε, ολοκλήρωση, την περιφερειακή, όταν είναι τέσσερις χώρες που υπέγραψαν και πολύ περισσότερες αυτές που δεν υπέγραψαν. Τι γίνεται με τις άλλες χώρες, λοιπόν, τώρα που έχουν υπογράψει αυτές οι τέσσερις χώρες τις διάμεσες συμφωνίες, τι γίνεται με τις υπόλοιπες που δεν έχουν υπογράψει η επίπτωση ποια θα είναι. Τελικά μήπως είμαστε με το διέρη και βασίλευε, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Έπειτα, από τα στοιχεία που έχω εγώ για την Μαδαγασκάρη τουλάχιστον, ο ρυθμός της ελευθέρωσης πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Την πρώτη χρονιά για το 2030, 35% των εισαγωγών της αποφάσισε να ελευθερώσει και θα ανέβει στο 81% σε 50 χρόνια. Τα στοιχεία για τις άλλες χώρες δεν τα ξέρω και τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά στην εσωτερική οικονομία. Τι συνέπειες ε, θα έχουμε στην ασφάλεια τροφίμων. Οι πρέσβεις, οι πρεσβείες έχουν κάποια άποψη επίσης για τη στάση των συνδικάτων, των οργανώσεων, των γεωργών, για τον αντίκτυπο που έχουν οι συμφωνίες αυτές επιτόπου. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να ελέγξει το 80% από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι φτάνει στο 95% για τι ε, Σεχέλε, αλλά εγώ φοβάμαι ότι με αυτόν τον τρόπο καταστρέφονται οι οικονομίε και κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από την ανάπτυξη και την αηφόρα ανάπτυξη. Η πραγματική φύση όλων αυτών είναι ότι στις ενδιάμεσε συμφωνίε δεν υπάρχει κανένα κεφάλαιο για την αηφόρα ανάπτυξη, δεν υπάρχει ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε η πραγματικότητα ε, τελικά είναι διαφορετική από αυτά που ακούμε και αυτά είναι που πρέπει να προσέξουμε πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχω κανέναν άλλον που να θέλει να ρωτήσει κάτι. Συνεπώς. Α, ο κύριος Κάσπαρη. Ναι. Παρακαλώ. Ο συνάδελφός μου που μίλησε πριν από μένα ανέπτυξε κάποιες συγκεκριμένες επιφυλάξεις βρίσκω ενδιαφέρον που και ευρωβουλευτής εκφράζει επιφυλάξεις αλλά και από τους εκπροσώπους των χωρών που προσήλθαν και που είπαν ότι υπερτερούν οι θετικές πτυχές. Αν μπορούσαν οι εκπρόσωποι να μας εξηγήσουν πώς βλέπουν τις επιφυλάξεις του συναδέλφου μου που μίλησε πριν. Πρόκειται στις περισσότερες περιπτώσεις τουλάχιστον για δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις των χωρών σας θα ήθελα λοιπόν να με πληροφορήσετε πώς βλέπετε την κατάσταση εσείς επιτόπου στις χώρες σας. Ο Πρόεδρος. Και εγώ πιστεύω ότι οι καλύτεροι κριτές των συμφωνιών μας είναι οι ίδιοι οι αντισημερώμενοι μας. Οι ίδιοι. Εσείς εκπροσωπείτε το λαό της Ζιμπάμπουε. Όχι. Ούτε και σε εκπροσωπεί το λαό της Ευρώπης. Οι Ζιμπαμπουανοί και οι Μαυριτιανοί είναι εδώ. Ας αποφασίσουν οι ίδιοι. Ανεξάρτητα και αυτόνομα. Αντί να προσπαθούμε να τους υποκαθιστούμε για το ποιο είναι το συμφέρον τους. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Ανέκυψαν ένα-δύο σημεία που ίσως θα πρέπει να επαναληφθούν. Ε, και θα πρέπει να επαναλάβω και κάποια από αυτά που είπα πριν. Για την περίφημο κανονισμό για πρόσβαση στην αγορά. Είναι ευπρόσδεκτο το ότι οι τέσσερις παρούσες χώρες χρησιμοποίησαν τον κανονισμό για πρόσβαση στην αγορά για το σκοπό που σχεδιάστηκε μετά από του 2008 μέχρι ότου έχουν επικυρώσει ή προσωρινά έχουν φάσει τη συμφωνία να γεφυρώσουν το κενό. Και αυτό συνέβη. Και χαιρόμαστε που το έκαναν αυτό. Ε, ντροπή που δεν το κάναμε αυτό με κάποιες από τις άλλες χώρες. Εφαρμόστηκε προσωρινά μόνο από τον Μάιο. Είμαστε στα πρώτα στάδια αλλά στα πλαίσια του κανονισμού για πρόσβαση στην αγορά πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκ των προτέρων έδωσε πρόσβαση ε, αδασμολόγητη σε αυτές κατά κάποιο τρόπο εφαρμόζαμε τη συμφωνία σε αυτούς από 1η Πρώτου 2008. Ε, αυτό συμπεριλαμβάνει ε, βελτιωμένους κανόνες ε, προέλευσης κλπ. Από την πλευρά μας μεν ήμασταν παρόντες, αλλά είναι σαφές ότι για τις χώρες, τις εμπλεκόμενες, ξεκίνησαν μόλις 1η Μαΐου ή τον Μάιο και είμαστε στην αρχική φάση δημιουργίας θεσμών πρέπει να το λάβουμε υπόψη και θα βρούμε βήμα για διάλογο στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας στι 19 Δεκάτου. Όσον αφορά το μέλλον, ε, ο κύριος Μέρφυ αναφέρθηκε στις πτυχές περιφερειακής ολοκλήρωσης. Εγώ τι έλεγα. Πρώτα απ' όλα είναι πρόσδεκτο το ότι οι τέσσερις χώρες μπόρεσαν να συνεργαστούν για να επιτευχθεί συμφωνία. Δεν είπα τίποτα περισσότερο είναι ένα βήμα προς την περιφερειακή ολοκλήρωση. Θα ήλπιζα και θα προσέβλεπα σε μια διαδοχική συμφωνία η οποία θα είναι περιφερειακή και θα σε περισσότερες χώρες από ό,τι παρούσα, αλλά πάντα θα υπάρχει κάποια διαφορά, ένταση μεταξύ της προθυμίας, της βούλησης για περιφερειακή ολοκλήρωση από τη μια και το επίπεδο φιλοδοξής συμφωνίας από την άλλη. Και γι' αυτό, πάνω σε αυτό θέλαμε να είμαστε ρεαλιστές και ευέλικτοι, ούτω ώστε θέματα όπως οι υπηρεσίες ή οι δημόσιες προμήθειες που δημιουργούν δυσκολίες σε κάποιες χώρες να συμπεριληφθούν σταδιακά και να μην επιβληθούν από την ε, πρώτη μέρα. Έγινε λόγος για αναπτυξιακή συνεργασία. Ε, αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε στις συνεδρίες επόμενης εβδομάδας. Προσβλέπουμε σε αυτό. Δεν θα αναφερθώ σε αυτό τώρα. Ε, θα ήθελα να πω ότι μπήκαμε στο όλο εγχείρημα με ανοιχτό πνεύμα και προσβλέπουμε σε συνέχιση της εφαρμογής της παρούς συμφωνίας και στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις που θα εκτηριχθούν σε παρόν πνεύμα. Ευχαριστώ πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή για τελική ε, παρέμβαση. Ε, ήθελα να ρωτήσω τους φιλοξενούμενους μας αν ήθελαν να κάνουν κάποιο σύντομο σχόλιο. Η κυρία Πρέσβυρα, έχετε το λόγο. Για δύο λεπτά ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναφερθώ σε δύο σημεία. Όσον αφορά την περιφερειακή φύση, σας διαβεβαιώνω ότι εμείς οι χώρες της Ανατολικής ε, και Νότιας Αφρικής συνεχίζουμε τις συζητήσεις για την ΕΠΑ. Την τελευταία εβδομάδα μαζί με τις υπόλοιπες χώρες ε, ε, ΕΣΑ στη Λουζάκα συζητήσαμε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά υπάρχει κάποια παρεξήγηση μεταξύ μας. Έχουμε στην ε, ΕΣΑ και χώρες που έχουν προτιμη, προτιμησιακή αντιμετώπιση που έχουν και άλλες δυνατότητες πρόσβασης. Αυτές που δεν ανήκουν εκεί πρέπει να προσπαθήσουν να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Δεν κάναμε κάτι πίσω από τις πλάτες των εταίρων μας. Ανοιχτά κινηθήκαμε. Η ΕΣΑ δέχεται αυτή την ανάπτυξη, θεωρεί ότι είναι μια κίνηση από την οποία μπορούμε να μάθουμε και θα συμπεριληφθεί στις γενικές διαπραγματεύσεις για ΕΠΑ. Όσον αφορά την αντίθεση του κοινού για τα στοιχεία για απελευθέρωση των αγορών, δεν σας έδωσα στοιχεία, αλλά έμεσα αναφέρθηκα για το Ζιμπάμπουε. Είμαστε δεσμευμένοι να απελευθερώσουμε τι αγορέ. Θέλουμε αμφίδρομη όμω ε, συνεργασία για την απελευθέρωση. Από τη μία θέλουμε να ενισχυθεί η βιομηχανία μα για να ανοίξουμε σταδιακά στους Ευρωπαίους εταίρους. Δεν μπορούμε ότι ανοίγουμε, γκρεμίζουμε τα τείχη 80% σε μια μέρα όταν δεν μπορούμε να εμπορευτούμε μαζί σας. για την αντίδραση του κόσμου. Νομίζω ότι είπα ότι το κοινό μαζί με τις εταιρείε λένε το εξής. Εάν δεν συμπεριληφθεί η αναπτυξιακή συνιστόσα στην αρχή της εφαρμογής της ΕΣΑ θα έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ήμουν παρούσα στις τελευταίες διαπραγματεύσεις ΕΠΑ στο Αράλε συζητήθηκαν τεχνικά θέματα. Εκπροσωπεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έγιναν δηλώσεις από εκπροσώπους τη Βιομηχανία που αυτό έλεγαν. Η βιομηχανία θα ήθελα να συμμετάσχει, αλλά θέλει να συμμετάσχει επί μιας δίκαιης, ισότιμης ε, βάσης. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λε Πρόεδρος. Ε, η Ζιμπάμπουε. Α, συγγνώμη. Η Μαδαγασκάρη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταλαβαίνω απόλυτα τους δύο βουλευτές που εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τις θετικές μας τους υπήν και διακηρύξεις. Τι είπαμε εδώ, υπενθυμίσαμε το πνεύμα που μας, το οποίο επικρατεί στις ε, διαπραγματεύσεις και στο οποίο κινούμεθα δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Πριν έρθουμε να διαπραγματευτούμε του Ευρωπαίου εταίρου, είναι προφανέ ότι επιτόπου ε, ερχόμαστε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Ε, μας δίνουν μια εντολή, ερχόμαστε με εντολή και η ανησυχία, της, η των κοινωνία των πολιτών, των συνδικάτων, των αγροτών μας την υπόψη την εντολή που μας δίδεται για να διαπραγματευτούμε. Για τη Μαδαγασκάρη, για τη συγκεκριμένη περίπτωση Μαδαγασκάρης, στις διαπραγματεύσεις ε, για την ε, διάμεση συμφωνία μπορέσαμε να πετύχουμε το εξής 20% των ευαισθητών όπως αποκαλούνται προϊόντα, προϊόντων να εξαιρεθούν από την απελευθέρωση. 20%. Ε, δεν είναι και άσχημα. Ε, σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι τα συμφωνία συμφέροντα της εσωτερικής μας οικονομίας δεν πλήττονται από την συμφωνία αυτή, λαμβάνονται υπόψη και τα συμφέροντα της κοινωνίας των πολιτών εν γέννη. Και κλείνοντας, θα ήθελα να επιβεβαιώσω κάτι για μας, τις αφρικανικές χώρες, η περιφερειακή ολοκλήρωση είναι ζωτική σημασία. Είναι σημαντικότατη για μας και στις διαπραγματεύσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα φροντίσουμε ούτω ώστε οι συμφωνίες αυτές να μην υπονομεύουν την διαδικασία ε, περιφερειακής ολοκλήρωσης που λαμβάνει η χώρα στην ε, Αφρική. Αυτό συνεχώς το έχουμε υπόψη. Και σας διαβεβαιώνω, διαβεβαιώνω τους παρόντες βουλευτές γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ε, εν τέλει ο Μαυρίκιος, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ και εκείνους που πήραν το λόγο και έθεσαν ερωτήσεις. Να πω απαντώντας όσον αφορά τις συνέπειες της ε, απελευθέρωσης που έθιξε ένας βουλευτής η απελευθέρωση πάντα ήταν και είναι επώδυνη διαδικασία κυρίως για μικρές αναπτυσσόμενες χώρες όπως είναι ο Μαυρίκιος συνεπάγεται κοινωνικό κόστος και οικονομικό κόστος όσον αφορά το κοινωνικό κόστος βλέπουμε στη διαδικασία μας της απελευθέρωσης για την οποία δεσμευτήκαμε πριν από χρόνια έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές απολύσει σε κάποιε μηχανίε και κλείσιμο εργοστασίων. Ε, πολλά κλείσιματα εργοστασίων που είχαν αρνητικέ συνέπειε. Και τα συνδικάτα εξέφρασαν ε, πάνω σε αυτό ανησυχίε. Όμω, απ' την άλλη, όπω είπαν και άλλοι ομιλητέ τη ομάδα μα, είμαστε δεσμευμένοι να ακολουθήσουμε την διαδικασία και θέλουμε να δώσουμε θελτικό μήνυμα προ τον κόσμο ότι θέλουμε να συμμορφωθούμε στου περιφερειακού κανόνε και στου παγκόσμιου κανόνε για το εμπόριο και γι' αυτό προχωρούμε στι διαπραγματεύσει αλλά, αλλά όπως προαναφέραμε για να ακολουθήσουμε το δρόμο της απελευθέρωσης χρειάζομαστε βοήθεια και στήριξη ούτως ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τουλάχιστον ε, την απε, τις της απελευθέρωσης να προστατεύσουμε τους στοχούς το λαό γι' αυτό ζητάμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας δώσει βοήθεια για το κόστος που πρέπει να καταβάλουμε για την προσαρμογή στα μέτρα που απαιτούνται για να ακολουθηθεί η διαδικασία της απελευθέρωσης. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο Κάσπαρη, τελευταίες παρατηρήσεις. Για, από τη δική μου πλευρά, ευχαριστίες και στην Κομισιόν για τις εξηγήσεις, αλλά και στους εκπροσώπους των συμβαλωμένων χωρών που μας εξήγησαν ποιες είναι οι δικές τους θέσεις και λυπούμε πολύ που ο συνάδελφο που μίλησε προηγουμένω εξήλθε τι αιθούσει και δεν άκουσε τι απαντήσει. Ή δυνατόν θα υποβάλω το σχέδιο εκθέσεως μου τον Νοέμβριο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα με την επεξεργασία του φακέλου αυτού. Βεβαίω είμαι στη διάθεσή σα για οτιδήποτε με χρειαστείτε. Πρόεδρο ευχαριστώ πολύ. Εξέταση του σχεδίου εκθέσεως στις 27 Νοεμβρίου και 28. Κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε άλλα θέματα σήμερα. Ευχαριστώ και η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 6 ε, Νοεμβρίου 9 το πρωί.